Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε λοιπόν με αυτήν την σημαντική κοινοβουλευτική στιγμή. Μια σημαντική στιγμή της θητείας μας που είναι η ακρόαση όσον αφορά την οριστήσα επίτροπο, την κυρία Ούλβα Γιωχάνσον. Καλώς ήρθατε εδώ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελευθεριών του Πολίτη. Καλώς ήρθατε, ναι. Θερμό χειροκρότημα. Θέλω να σας θυμίσω λιγάκι τη διαδικασία. Πρώτον, σύμφωνα με το παράρτημα 7 του κανονισμού που περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει τους οριστέντες επιτρόπους βάσει των γενικών τους ικανοτήτων, των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν και την ανεξαρτησία τους. Στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε την γνώση όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσωτερικών υποθέσεων όπως επίσης και τις ικανότητες επικοινωνίας. Σας επιθυμίζω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε διάφορες ερωτήσεις στην οριστήσα επίτροπο με δύο κοινέ ερωτήσεις από κοινού την διάσκεψη των Προέδρων και άλλες που προετοίμασε η Επιτροπή μας. Η οριστήσα Επίτροπος έχει διαπαντήσει γραπτά. Οι ερωτήσεις αυτές και οι απαντήσεις έχουν διανεμηθεί στους ευρωβουλευτές της κοινοβουλευτικής αυτής επιτροπής σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω επίσης ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, δεν εξέφρασε ένσταση όσον αφορά τη διεξαγωγή της ακρόασης αυτής με την Οριστή επίτροπο Ούλβα Γιωχάνσον. Συνεπώς, η συζήτηση θα διαρθρωθεί ως εξής. Πρώτον, η οριστή επίτροπος θα παρουσιάσει τα θέματά της με μια αρχική παρουσίαση 15 λεπτών το πολύ. Και στη συνέχεια, αμέσως μετά, θα υπάρξουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Το πολύ 25 ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. Όσοι ήθιστε, θα αρχίσουμε με ερωτήσεις αναπολιτική ομάδα, σύμφωνα με την σταθμισμένη δύναμη της κάθε πολιτικής ομάδας βάσει του συστήματος Χόντο. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Λοιπόν, οι ερωτήσεις θα είναι πέντε λεπτά, ένα λεπτό η ερώτηση από τον Ευρωβουλευτή, δύο λεπτά απάντηση. Και υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει αμέσως αντίδραση από τον Ευρωβουλευτό για άλλο ένα λεπτό από τον ίδιο Ευρωβουλευτή έτσι που υπέβαλε την ερώτηση και ένα λεπτό μια δεύτερη απάντηση από την οριστή σε επίτροπο. Και αυτό ζητάμε το σύστημα να ακολουθήσουν οι πρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Και μετά θα έχουμε και δεύτερο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων με όλες τις πολιτικές ομάδες, αλλά και με εκπροσώπους των μη εγγεγραμμένων, κάποιους από τους μη εγγεγραμμένους δηλαδή. Και στο τέλος της ακροάσεως η οριστής επίτροπος θα έχει και 5 λεπτά στη διάθεσή της για το κλείσιμο. Μην ξεπερνάτε το χρόνο σας παρακαλώ. Να το έχετε υπόψη σας αυτό, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο χρόνος θα τηρείται πλήρως. Αλλιώς... Θα αναγκαστώ να διακόπτω. Να σας ζητάω να ολοκληρώνετε ή να σας κόψω το λόγο στο τέλος και δεν θα ήθελα εδώ να κόψω το λόγο σε κανέναν. Γι' αυτό να είσαστε συνεργάσιμοι παρακαλώ και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόησή σας. Έχουμε διερμηνία στην ακρόαση αυτή σε όλες και τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην μιλάτε λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα σας παρακαλώ, ώστε να μπορέσουν τα συστήματα και διερμηνείς να μεταφράσουν αυτά που λέτε. Η συζήτηση επίσης μεταδίδεται στο διαδίκτυο στο, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορείτε να έχετε και μετά πρόσβαση στις μακροσκοπημένες ακροάσεις στην ίδια στο σελίδα. Αυτά και τα προκαταρτικά. Τώρα, η ακρόαση αυτή πρέπει να ξέρουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την Επιτροπή μας. Πρώτα απ' όλα γιατί θα είναι η μόνη ακρόαση ε, στην οποία είμαστε η αρμόδια υπεύθυνη Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δηλαδή που δεν οργανώνουμε την ακρόαση αυτή αποκινούμε κάποια άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Είμαστε μόνοι μας εδώ, κυρίως όταν πρόκειται για την ομοθεσία στα θέματα ε, τα σχετικά με αυτό το χαρτοφυλάκιο, βάσει της συνθήκη της Λισαβόνας, εμείς είμαστε αρμόδιοι για την πολιτική ασύλου και μετανάστευση, για την διαχείριση των συνόρων και τις σχετικές πολιτικές, αλλά επίσης και, και αυτό είναι σημαντικό, για την πολιτική εσωτερικής ασφάλειας, πολέμηση δηλαδή του οργανωμένου εγκλήματος, του διασυνοριακού εγκλήματος, της Τρομοκρατία. Και επίση είμαστε υπεύθυνοι για τα περί Ευρωπαίου εισαγγελέα. Συνεπώς, θα ανταλλάξουμε απόψει για όλα αυτά τα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής που έχουμε μπροστά μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα τελευταία χρόνια όπως έχουμε δει. Αρχίζουμε λοιπόν ευθύ αμέσω και δίνω το λόγο στην κυρία Ιούλβα Γιωχάνσον για να μας κάνει την παρουσίασή της. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για τα επόμενα 15 λεπτά παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ ενώπιον, ενώπιον σας. Ε, καταλαβαίνω ότι θα μου κάνετε τη ζωή λίγο δύσκολη, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι παρότι έχω τρακ, ε, περίμενα τη στιγμή αυτή, διότι είναι μια ε, βασική στιγμή της δημοκρατίας και είσαστε οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Είσαστε οι άνθρωποι που πρέπει να οργανώσετε την ακρόαση αυτή και να ε, αποφασίσετε αν μπορώ να αναλάβω τα καθήκοντά μου ως Επίτροπος. Ε, και προσλέπω λοιπόν στη συζήτηση αυτή και προσλέπω, ε, ελπίζω, και στη συνεργασία μαζί σας τα επόμενα πέντε χρόνια. Ήμουνα υπουργό σε πέντε διαφορετικέ κυβερνήσει τη Σουηδία με τρει διαφορετικού πρωθυπουργού. Ήταν όλε κυβερνήσει μειοψηφία. Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει η στενή συνεργασία ανάμεσα σε διάφορες πολιτικές ομάδες και η εξέβρεση συμβιβασμών ε, με το Κοινοβούλιο. Και Καταλαβαίνω ότι θα χρειαστώ και εδώ τις ε, εμπειρίες μου αυτές. Το 2015 η Σουηδία ε, υποδέχτηκε περισσότερους πρόσφυγες κατά κεφαλήν από ότι οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Το 1 τρίτο όλων των ασυνόδευτων ενηλίκων που κατέφτασαν στην Ευρώπη έφτασαν ε, στη Σουηδία. Ήταν μεγάλη πρόκληση. Ο Πρωθυπουργό μου ανέθεσε την ειδική ευθύνη να συντενίσω όλες τις ενέργειες της κυβέρνησης που είχαν να κάνουν με την μετανάστευση και την ενσωμάτωση στην κοινωνία της Σουηδίας. Είμαι περήφανη που η Σουηδία μπόρεσε να ε, αποτελέσει καταφύγιο για τόσους πρόσφυγες στο χρονικό αυτό διάστημα και που τόσοι από αυτούς τώρα πια έχουν ενταχθεί στη σουηδική κοινωνία και συμβάλλουν στην ε, ανάπτυξη της οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως ε, κατά το διάστημα αυτό συνειδητοποίησα ότι μας λείπει ένα λειτουργικό και διαχειρίσιμο ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης και ασύλου. Πραγματικά χρειαζόμαστε κοινέ και βιώσιμες ευρωπαϊκές λύσεις στη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε λύσεις που να επιτρέπουν ε, τον προγραμματισμό και ε, στα άτομα και στην κοινωνία. Οι πολιτικές ε, μετανάστευσης και ασφαλείας είναι σημαντικές και είναι, ενισχύουν αμοιβαία μία την άλλη, είναι όμως ξεχωριστές. Η μετανάστευση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απειλή στην ασφάλεια. Η ασφάλεια συνδέεται με την ελευθερία. Όλοι στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ζουν σε μια κοινωνία σύμφωνα με, όπου να επικρατεί το κράτος δικαίου, έχοντας ε, τη συνείδηση ότι οι δημόσιες αρχές κάνουν ό,τι ε, μπορούν για να τους προστατεύσουν και να ε, ε, καταπολεμήσει αυτούς που διακυβεύουν την ελευθερία αυτή. Οι απειλές στην ελευθερία είναι απειλές στις κοινωνίες μας. Πρέπει όμως να πω επίσης ότι θα επαγρυπνώ ώστε να διασφαλίσω οι ελευθερίες που θέλουμε να προστατεύσουμε να μην διακυβεύονται από τα μέτρα ασφαλείας. Όσον αφορά τη μετανάστευση, αποστολή μου είναι να βρω έναν νέο τρόπο που να λειτουργεί και που να είναι πιστός στις αξίες μας. Η βασική μου ε, προτεραιότητα, και θα είναι δύσκολο αυτό το καταλαβαίνω, είναι να αναπτύξω το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Θα είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει όμως επίσης να καταστήσω σαφές ότι δεν μας παίρνει να αποτύχουμε. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Έχουμε προχωρήσει πολύ, έχουμε καταφέρει πολλά, αλλά παραμένουν κάποιες ε, πολύπλοκες προκλήσεις. Τώρα λοιπόν έχει δοθεί θετική ορμή για να τις αντιμετωπίσουμε με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που να χτίζει γέφυρες και όχι τύχη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η ασφάλεια και η μετανάστευση αποτελούν προτεραιότητες στις πολιτικές κατευθυντήρες γραμμές διότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στους πολίτες στα θέματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Και η μετανάστευση και η ασφάλεια είναι από τις τρεις κορυφαίες προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Η ασφάλεια και η μετανάστευση ε, αφορούν, ε, σχετίζονται με πολλές πολιτικές εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ο συντονισμός είναι υψίστης τη σημασίας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση και να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να ε, πετύχουμε συμβιβασμούς και συνεργασία που είναι ε, η θεμελιώδης λύθη του ευρωπαϊκού τρόπου συνεργασίας. Και έτσι σκοπεύω να προχωρήσω. Γνωρίζω ότι εσείς ως ευρωβουλευτές και ως μέλη αυτής της σημαντικής επιτροπής ε, έχετε πολλές γνώσεις και πείρα πάνω σε αυτόν τον τρόπο εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αξίες και αυτές θα πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες αρχές μας όχι μόνο θα υπερασπιστώ ε, και τις αξίες αυτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και απέναντι στο υπόλοιπο του κόσμου. Για μένα είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τις δημοκρατίες μας από τον λαϊκισμό και τον εξτρεμισμό και πάντα να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει να αντιμετωπίσω τις σημαντικές προκλήσεις ε, στις ε, εσωτερικές υποθέσεις. Ε, δεν θα προτιμούσα άλλο χαρτοφυλάκιο. Αυτό ακριβώς προτιμούσα και ε, είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ε, η εκλεγήσα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνοντάς μου τόση εμπιστοσύνη. Οι απειλέ που αντιμετωπίζουμε στον, τόπο, στον τομέα τη ασφάλεια, εξελίσσονται συνεχώ και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε τα κενά στην προσέγγιση ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εσωτερική της ασφάλεια. Ε, Στόχο μου είναι να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική ένωση ασφαλεία που να βασίζεται στα θεμέλια που έχουν ε, τεθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι αποτελεσματική η νομοθεσία, να εφαρμόζεται και θα πρέπει να κλείσουμε τα κενά στο πλαίσιο ασφαλείας μας. Το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, η διακίνηση ανθρώπων, ε, η εμπορία ανθρώπων και η ε, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ε, αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για μένα. Συνήθω ε, τα θύματα είναι τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας ε, και η κοινωνία μα θα πρέπει να του προστατεύσει. Εγώ λοιπόν θα του υπερασπιστώ, θα εργαστώ ακούραστα για να ε, κλείσω, να περιορίσω το, δυνατό χώρο για τους τρομοκράτες να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τις επιθέσεις τους. Θα καταπολεμήσω επίσης κάθε μορφή ριζοσπαστικοποίησης. Θα ήθελα να επενέσω την έκθεση της Επιτροπής ΤΕΡ. Οι συστάσεις αυτές θα με κατευθύνουν στι εργασίες μου πολύ σημαντικό για να πετύχουμε καλό αντίκτυπο είναι η καλύτερη συνεργασία όσον αφορά την επιβολή του νόμου. Πόσο μάλλον ε, με τις ε, ε, ραγδαίε εξελίξεις που βλέπουμε όσον αφορά τις νέες απειλές. Και η Europol θα πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο. Θέλω μία προσέγγιση που να βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία και στόχος μου είναι να εφαρμόσω τις αρχές της καλύτερης νομοθεσίας ε, όσον αφορά την ε, εκπόνηση μελλοντικών ε, προτάσεων στο χαρτοφυλάκιο μου. Όσον αφορά την μετανάστευση, όπως όλοι γνωρίζετε, οι συζητήσεις αυτές ήταν δύσκολες και έχουν οδηγήσει σε διχασμό. Υπάρχει επίγους ανάγκη για κοινέ, διαχειρίσιμες, βιώσιμες και προβλέψιμες λύσεις. Αυτή τη στιγμή ε, έχει δοθεί ορμή στα θέματα αυτά. Υπάρχει νέα κίνηση με την άφηξη της ε, Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και έχω λάβει σαφή εντολή από την σαν Πρόεδρο να προτείνω ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης και σύλλου. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσω προσεκτικά τις διάφορες απόψεις για να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινά στοιχεία. Με το Κοινοβούλιο φυσικά, αλλά και διμερώς με όλα τα κράτη-μέλη μόλις αναλάβω τα καθήκοντά μου, εφόσον εσείς εγκρίνετε τον διορισμό μου, ε, σκοπεύω να έχω πολύ γρήγορα διμερεί συναντήσει με όλα τα κράτη-μέλη και θα κρατήσω ενημέρη την Επιτροπή σας θα εξετάσω μία σειρά πολιτικών ε, μετανάστευσης για το άσυλο, την καταπολέμηση της ε, παράτυπης μετανάστευσης, ε, την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, την επιστροφή νόμιμες οδούς μετανάστευσης, ένταξη στην κοινωνία και συνεργασία με εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τμήμα αυτή της ολιστικής προσέγγισης θα είναι να εξετάσουμε προσεκτικά υπάρχουσες προτάσεις που έχουν ήδη τεθεί και είναι σημαντικό για μένα να έχουμε ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις μας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η Επιτροπή σας έχει εργαστεί πολύ σκληρά, ε, με ευρωπαϊκό τρόπο θα έλεγα, για να καθορίσει την αρχική της θέση πάνω σε πολλά από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας στον τομέα του ασύλου. Αυτή είναι σημαντική δουλειά, αυτή η δουλειά που έχει γίνει, πάνω στην οποία θα πρέπει να βασιστούμε θα πρέπει ε, καθοδηγητής μας ε, να είναι η επιθυμία για εξέβρεση βιώσιμων λύσεων. Πάντα προσπαθώ να βρω τρόπο να κλείσουμε τα παραθυράκια, ε, που, τα κενά που βρίσκονται ανάμεσα στο άσυλο και την επιστροφή. Ενώ πρέπει να μείνουμε πιστοί στις αξίες μας και τις διεθνείς μας ευθύνες, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε... Η όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέφουν. Πέρσι μόνο το 1 τρίτο όσων έλαβαν εντολή επιστροφής τελικά επέστρεψαν. Μια ένα αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα ασύλου χρειάζεται και μια λειτουργική και ανθρώπινη πολιτική επιστροφή σε που να σέβεται απόλυτα την αρχή ε, της μη επαναπρόθεσης του διεθνούς δικαίου. Οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές επίσης ετώνησαν την ανάγκη για νόμιμες και ασφαλές οδούς ε, μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει τμήμα της λύσης. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που το μερίδιο της Ευρώπης ε, στην διεθνή επανεγκατάσταση ανερχόταν ε, ε, στο 15% ε, στο 50% θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τις επίγουσες ανάγκες. Δεν μπορούμε επίσης να ανεχτούμε να κινδυνεύουν και να χάνονται ζωές στη Μεσόγειο. Ε, ζωτικό στοιχείο του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου θα είναι μια πιο βιώσιμη και αξιόπιστη και μόνιμη προσέγγιση ε, στην ε, αναζήτηση και διάσωση. Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τις ad hoc λύσεις τις, με μόνιμες λύσεις. Θα είναι ηθικό καθήκον μας να σώσουμε ζωές. Θα πρέπει επίσης να διαλύσουμε τις ε, εγκληματικές ε, συμμορίες ε, που διακινούν ανθρώπους. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ένα από τα επιτέρματα κλειδιά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο χώρος Σέγγεν. Βασικός μου στόχος, λοιπόν, θα είναι η γρήγορη επιστροφή σε έναν απόλυτα λειτουργικό χώρο Σέγγεν. Όσο πιο αποτελεσματικό ε, είναι το νέο σύμφωνο, τόσο πιο ισχυρά θα είναι τα εξωτερικά μας σύνορα ε, και ε, θα μας βοηθήσει η Frontex σε αυτό. Ενώ όσο πιο αποτελεσματική είναι η δουλειά μας κατά της εμπορίας ανθρώπων, τόσο πιο πολύ εμπιστοσύνη θα χαίρει ο χώρος Σέγγεν. Και έτσι θα μπορέσουμε να διευρύνουμε κιόλας τη ζώνη Σέγγεν. Στόχος ε, λοιπόν ε, είναι να έχουμε μια πολιτική ισορροπημένη και δίκαιη που να βασίζεται στις αξίες μας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο το χαρτοφυλάκιο αυτό. Αυτό μου λένε όλοι αυτές τις ε, τελευταίες τρεις εβδομάδες από τότε που ορίστηκα επίτροπος. Θα πρέπει όμως να προοδεύσουμε στον τομέα αυτόν. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτή λοιπόν θα είναι η ε, κορυφαία προτεραιότητά μου και θα χρειαστώ τη βοήθειά σας, την εμπειρογνωμοσύνη σας και την πείρα σας στον τομέα αυτόν. Είναι λοιπόν μεγάλη τιμή για μένα, θα είναι μεγάλη τιμή για μένα εάν εγκρίνετε τον διορισμό μου και προσβλέπω ε, στην ε, συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την σε Επίτροπο για την παρουσίαση αυτή. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές και θα αρχίσουμε με τους συντονιστές, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Αρχίζουμε, έχω εδώ τον κατάλογο των ομιλητών. Ε, μην ξεχνάτε, δύο λεπτά η ερώτηση, μετά ακούμε την απάντηση, μετά ένα λεπτό ακόμα ο Ευρωβουλευτής και ένα λεπτό η δεύτερη απάντηση. Αρχίζουμε με τον κύριο Τόμα Στόμπε, εκπρόσωπο του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε την υποψήφια επίτροπο. Χαίρομαι που μίλησε για πράσπιση των κοινών ευρωπαϊκών μας αξιών. Ελπίζω ότι αυτό σημαίνει ότι η υποψήφια επίτροπος θα υποστηρίξει επίσης και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ερώτηση. Κοινή ασφάλεια, ευρωπαϊκή ασφάλεια, πολιτική ασφάλειας Έχουμε τεράστια προβλήματα με όπλα, με ναρκωτικά που διασχίζουν τα σύνορά μας. Βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσει όσον αφορά τα εγκλήματα κατεδειχθησίας με κινητές ομάδες εγκληματικές που διατρέχουν την Ευρώπη. Λοιπόν, η ερώτηση, ποια συγκεκριμένα βήματα είσαστε έτοιμοι να κάνετε υποψήφια επίτροπε. Θα κάνετε περισσότερα, θα αυξήσετε τα κονδύλια για τη Europol. Είστε πρόθυμοι να εξασφαλίσετε ότι θα έχουμε ένα κέντρο που, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που στρέφεται κάτι της διοκτησίας. Έχετε το λόγο, κυρία Γιωχάντσον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Τομπέ. Είναι κρίσιμη σημασία να υπερασπιστούμε τις κοινέ μας αξίες. Να πω κάτι γι' αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Σημαντικές αξίες επί των οποίων βασίζεται η ένωσή μας απειλούνται απειλή Ξτρέφεται κατά του κράτους δικαίου, κατά των μειονοτήτων, υπάρχουν απειλές. Έχουμε ε, Εβραίους που για μία ακόμη φορά φοβούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δεν πρέπει να πανοχλούνται οι άνθρωποι, να υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Είναι ακρογωνίως λήθος για αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η προάσπιση αυτών των θεμελιωδών αξιών επί των οποίων βασιζόμαστε. Η ασφάλεια σχετίζεται με αυτά. Αν δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα σωστά, όπως είπατε κι εσείς, θα έχουμε προβλήματα με όπλα εκρηκτικά και ναρκωτικά που θα διέρχονται τα σύνορα. Και είναι κάτι που επηρεάζει τις κοινωνίες μας αυτό. Σαν δηλητήριο είναι αυτά. Όταν δεν μπορεί ο κόσμος να αισθάνεται ότι προστατεύεται σωστά από την κοινωνία, έναντι του εγκλήματος δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι οι οργανωμένοι εγκληματίε όλο και περισσότερο γίνονται πιο επαγγελματίε στα επιχειρηματικά μοντέλα που ακολουθούν και στου τρόπου του Και θα πρέπει να κινηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να του καταπολεμήσουμε σωστά. Όσον αφορά τα εγκλήματα κατά τη ιδιοκτησία είναι μία από τι προτεραιότητε που υφίστανται τώρα για τη Europol μαζί με τα κάτι μελη λήφθη απόφαση. Ήδη αποτελεί προτεραιότητα αυτό το ζήτημα που θίξατε. Ένα λεπτό για διευκρινιστική ερώτηση. Κάποια αντίδραση. Εκτός μικροφώνου, κ. Στομπέ. Ευχαριστώ, κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Κατανοώ ότι περασπίζεστε τις κοινέ μας ευρωπαϊκές αξίες. Θέλω μια διευκρίνηση όμως. Υποστηρίζετε και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής Εξίσου σημαντικό είναι μια υποψήφια επίτροπος να λέγει ότι είναι σημαντικό να αστιαστεί η Europol περισσότερο στα εγκλήματα κατά στιοκτησίας. Η ερώτησή μου αφορούσε περισσότερο κατά πόσο είστε πρόθυμοι και ανοιχτοί για συζήτηση, ώστε να εκτιμάσουμε, να δημιουργήσουμε ένα ειδικό κέντρο για την καταπολέμηση αυτού του φαινόμενου. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάθε κυβέρνηση και κάθε χώρα ξεχωριστά σε αυτή τη φάση. Για το θέμα ασφαλείας, ξέρω ότι προσπαθείτε να έχουμε ασφάλεια στα σύνορά μας. Θα ήταν ενδιαφέρον, έχετε χρόνο στην απάντησή σας, αν μπορείτε να δώσετε λεπτομέρειες. Τι θα κάνετε όσον αφορά την αύξηση της ασφαλείας στα σύνορά μας. Έχετε το λόγο κύριε Αποψήφια Επίτροπε. Ευχαριστώ λέει κύριε Γιώχανσον. Βέβαια υποστηρίζω τον Ευρωπαϊκό Τρόπο ζωή. Είναι κάτι που αφορά τις αξίες μας. Και είναι σημαντικότατο να προσπιστούμε αυτές τις αξίες. Αυτός είναι ευρωπαϊκός τρόπος ζωή θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ευρωπαϊκό τρόπο ζωή τη Ευρωπαϊκή μα Επιτροπή. Στον αφορά το έγκλημα κατά τη ιδιοκτησία και αν πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο γι' αυτό, δεν ξέρω. Δεν θα ήταν σοφό να απαντήσω συγκεκριμένα σήμερα. Δεν έχω λάβει ακόμα καθήκοντα. Α συνεχίσουμε το διάλογο περί επαρκούς χρηματοδοτήσεως της Europol και προτεραιοτήτων ε, τα επόμενα χρόνια για την Europol. Ευχαριστώ κύριε Γιωχάνσεν. Δεύτερος, ο συνάδελφος Κλοντ Μωράες. για ένα λεπτό. Κυρία Οριστής Επίτροπε, όπως είπατε, έχετε εμπειρία για τα θέματα αυτά. Την Κυριακή είδαμε φοβερές σκηνές στον καταβλισμό στη Μόρια. Και ξέρετε ότι το θέμα αυτό εδώ και χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και είναι θέμα του χαρτοφυλακίου σας. Είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε καλές πολιτικές. Γι' αυτό λέμε ότι είναι δύσκολο το χαρτόφυλλο σας. Πολλές φορές είπατε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να αποτύχουμε και ότι η αλληλεγγύη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το είπατε και το ξαναείπατε στην αρχική σας παρουσίαση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε Πλειοψηφίε για το Δουβλίνο, για τους διάφορους κανονισμούς. Τα καταφέραμε να πετύχουμε πλειοψηφίε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από, όλες, όλο το πολιτικό φάσμα το καταφέραμε αυτό. Το Συμβούλιο όμως κολλησιεργεί, δεν παίρνει τίποτα εκεί. Οπότε η ερώτησή μου είναι, εσείς τι θα κάνετε ώστε να επιτευχθεί πρόοδος αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Απάντηση κυρία Ιωάννσον. Σας ευχαριστώ κύριε Μωράες για την ε, όντω πολύ σημαντική αυτή ερώτησή σας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταφέρει με πραγματικά ευρωπαϊκό τρόπο να καταλήξει σε συμβιβασμούς για κοινή λύση. Όμως η κατάσταση έχει βρεθεί σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο εδώ και αρκετά χρόνια. Η αποστολή μου βέβαια είναι ακριβώς να βγάλω από τα αδιέξοδο αυτή την υπόθεση και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να το πετύχω αυτό. Πρώτα, όπως είπα, θα μιλήσω διμερώς με όλες τις χώρες μέλη για να καταφέρω να καταλάβω ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα, οι πιο σημαντικές συνιστώσεις όπου υπάρχουν οι διαφορές και μετά θα προχωρήσω. Από τη φύση μου δεν μπορώ να πω ότι έτσι θα γίνει, αλλιώς θα γίνει, γιατί ακριβώς αυτό θέλω. Να ακούσω πρώτα όλους του εμπλεκόμενου, όλες τις εμπλεκόμενε ε, πλευρές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια, που γνωρίζει καλά τα πράγματα, γιατί εσείς καταλήξατε στις συμφωνίες που καταλήξατε. Οπότε θέλω να τους ακούσω όλους. Μου έχει ανατεθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο και αυτή η αποστολή να πετύχω ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Και αυτό γιατί έχω εμπειρία στη διάθεσή μου, γιατί έχω ασχοληθεί με δύσκολα πράγματα. Έχω σπάσει πολλά αυγά στο παρελθόν στην πολιτική μου καριέρα. Και σίγουρα θα χρησιμοποιήσω πολλά μέσα για να το πετύχω και σίγουρα θα χρειαστώ τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως τη βοήθεια των έμπειρων μελών της Επιτροπής αυτής. Πιστεύω ότι είναι εφικτό. Αυτό. Πρόεδρος, εσείς κύριε Μωράες τώρα, για μια σύντομη αντίδραση. Αναγνωρίζω το θετικό τόνο της παρουσίασής σας, κυρία Οριστήσα Επίτροπος, αλλά αν ε, δεν τα καταφέρνουμε. Όντως, ε, το αδιέξοδο βρίσκεται στο Συμβούλιο. Αν εξακολουθήσει με το αδιέξοδο αυτό το Συμβούλιο, ρωτάω, τι θα κάνουμε. Υπάρχει η ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στη συνθήκη. Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να αλλάξει δηλαδή να προχωρήσουμε όντως στην απόφαση με ειδική πλειοψηφία αντί για την ομοφωνία στο Συμβούλιο. Αλλιώς φοβάμαι ότι θα ξαναβρεθούμε σε αδιέξοδο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Κυρία Γιωάνντσον. ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα είναι καλό να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε το σύμφωνο αυτό και για τη μετανάστευση και για το άσυλο, που σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερα πράγματα να συζητήσουμε στο τραπέζι. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε κοινό σημείο κίνηση. Τώρα, αν αναλάβω τα καθήκοντά μου την 1η Νοεμβρίου, θα αρχίσω να προσπαθώ ε, να πετύχω όσο ευρύτερο συμβιβασμό γίνεται. Αυτό είναι ο στόχος μου, ε, να καταφέρω να συμφωνήσουν όλοι. Στο τέλος, εννοείται ότι χρειαζόμαστε έτσι καλώς ένα νέο σύμφωνο. Ευχαριστώ εκπρόσωπος της ομάδα Renew τώρα, ο κύριος Σουντεράτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Οριστήσα Επίτροπε, ε, θα αναφερθώ στην περιοχή Σέγγεν που έγινε συνώνυμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ε, και αποτελεί μια από τις ε, σημαντικές επιτυχίες που μπορέσαμε να ε, παραδώσουμε στους πολίτες μας. Κάποια κράτη-μέλη ε, έχουν ε, επιβάλει ε, επιπλέον ελέγχους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί να το επιπλήξει αυτό το νομιμοποίησε. Και επίσης ε, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία έχουμε ανθρώπους που περιμένουν στο κατόφλι του Σέγγεν ε, χωρίς να υπάρχει κάποια απάντηση για το πώς ε, και πότε θα μπορέσουν να εισέλθουν. Εσείς είπατε ότι μια πλήρως λειτουργική περιοχή Σέγγεν θα αποτελέσει στοιχείο κλειδί του νέου συμφώνου, αλλά οι κανόνες ήδη τώρα παραβιάζονται. Συγκεκριμένα, Πώς και πότε θα διασφαλίσετε να μην χαθεί ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιωχάνσον, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Όπως είπα και κατά την εισαγωγή μου, η σύντομη επιστροφή σε μια πλήρως λειτουργική περιοχή Σέγγεν αποτελεί προτεραιότητα και αυτό αναφέρεται ε, και στην επιστολή ανάθεσης ε, καθηκόντων μου. Αυτό βέβαια θα απαιτήσει διάλογο με τα κράτη-μέλη που έχουν εισάγει εσωτερικούς ε, συνοριακούς ελέγχους. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε κιόλας ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα σε μια πλήρως λειτουργική περιοχή Σέγγεν και κάποια από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην δέσμη μέτρων για το άσυλο. Διότι οι ισχύοντες κανόνες του Δουβλίνου δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούν πολύ καλά. Αυτά λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους. Θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε. Συμφωνώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τουράτση, έχετε βάλει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να ε, θέτει κανείς ερωτήσεις με απάντηση ναι ή όχι, αλλά θα προσπαθήσω. Θα ξεκινήσετε διαδικασίες παραβάση απέναντι στα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν ε, τέτοιους εσωτερικούς νεριακούς ε, ελέγχους ε, εν αναμονή του νέου συμφώνου. Και επίσης τι χρονοδιάγραμμα δίνετε στον εαυτό σας απέναντι στο Συμβούλιο. Κύρια Γιωχάνσον, σας ευχαριστώ. Φυσικά. Ε, η ίστατη λύση είναι πάντα η διαδικασία επιπαραβάση. Αυτό είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό πάντα μπορεί να συμβεί. Νομίζω όμως ότι ε, αν αναλάβω τα καθήκοντά μου την 1η Νοεμβρίου, δεν θα πρέπει να ξεκινήσω από εκεί, θα πρέπει να ξεκινήσω από διάλογο με τα κράτη-μέλη και να προσπαθήσω να βρω λύσεις ε, προτού ε, προχωρήσουμε σε διαδικασίες επί παραβάση. Και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και πώς ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε στο θέμα αυτό, θα επανέλθω σε αυτό όταν θα έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου και θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε μαζί. Καλώς για τους πράσινους. Ο συνάδελφο, η κυρία Στρίκη, συνάδελφό μα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητή υποψήφια επίτροπε. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να εστιάζεται στην εξωτερική συνεργασία για τη μεταστατική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ενώ οι παρούσε πρακτικέ στην Τουρκία και στη Λιβύη δημιουργούν τεράστιε ανησυχίε. Η Τουρκία απειλεί να απελάσει ένα εκατομμύριο ε, πρόσφυγε. Να του επιστρέψει στη Συρία και πάτη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ενώσεω Τουρκία και τη συνεργασία με τη Λιβύη αυξάνεται ο κίνδυνος παραβίασης των δικαιωμάτων των μεταναστών, διότι ε, ξαναεπιστρέφουν σε φρικτές ε, συνθήκες. Μαζεύονται μάλλον σε φρικτές συνθήκες στη Λιβύη. Είπατε ότι θα δείτε πώς θα αξιολογήσετε και θα παρακολουθήσετε τον καλύτερο τρόπο τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλε τι μορφέ συνεργασία με τρίτε χώρε. Αυτό το επικροτούμε. Τι νέα βήματα όμω θα λάβετε για να πετύχετε αυτό συγκεκριμένα και πώ θα ενημερώνετε και θα εμπλέξετε και το κοινοβούλιο στη διαμορφώση αυτών των αποτελεσμάτων. Και θα είσαστε σίγουροι ότι αυτή η παρακολούθηση θα συμπεριλαμβάνει αναξιολόγηση διαφανή και ανεξάρτητη και θα διεξάγεται και θα μοιραστείτε μαζί μα αξιολόγηση συνεπειών πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξεκινήσει τέτοια συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε παραβίαση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχετε δύο λεπτά, κύριε Γιωχάνσο, την απάντησή σας. Απάντηση, ευχαριστώ πολύ, κυρία Στρίκ. Πολλές ερωτήσεις μου θέσατε. Να ξεκινήσω από το εξή. Η κατάσταση Λιβύη είναι φρικτή. Απέσια για του πρόσφυγες έχουν κολλήσει εκεί σε συνθήκε που κανένα ανθρώπινο όν δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει και να ζει σε αυτές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα συνεργάζονται με την ύπατη αρμοστία το ΟΗΕ και το IOM για να προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε αυτού του ανθρώπου από αυτή την αποτελμάτωση στη Λιβύη και εκεί μπορούμε να αναπτύξουμε αυτού του είδους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, να βοηθήσουμε τον κόσμο να φύγει από τη Λιβύη, να μετεγκατασταθεί σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να προχωρήσω. Βέβαια, πρέπει να βασιστώ στην προθυμία των κρατών μελών να υποδεχθούν τους μετεγκατασταθέντες μετανάστες θα έχουμε αύξηση του αριθμού των μεταγκαταστάσεων. Είχαμε τα τελευταία χρόνια αύξηση μεταγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία και ίσως ότι ο τρόπος μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει μπλοκαριστεί ε, στη Λιβύη σαν πρόσφυγας. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρίκ, κυρία Στρίκ, κοιτάξτε, ανέφερα τη Λιβύη και την Τουρκία σαν παραδείγματα Συνεργασία, που η συνεργασία τελικά βλάπτει τα δικαιώματα των μεταναστών. Αυτά ήταν τα παραδείγματα. Προσπαθούμε να μειώσουμε αυτή τη βλάβη η ερώτησή μου είναι η εξή. Πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά του δεν πλήττονται σαν αποτέλεσμα αυτή τη συνεργασία. Αν είστε σοβαροί στην απάντησή σα, στη γραπτή απάντηση ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών είναι βασικό στοιχείο τη εξωτερική πολιτική και μετανάστευση, είσαστε πρόθυμοι να πάρετε το πρώτο βήμα, δηλαδή να εξασφαλίσετε αξιολόγηση συνεπειών και ανεξάρτητο έλεγχο και εποπτεία Συμφωνείτε επίση ότι αυτό είναι απαραίτητο για να τηρήσετε την υπόσχεσή σα ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι βασική πτυχή. Εν τη αυτή περιπτώση μπορείτε να δεσμευτείτε πάνω σε αυτό και να μοιραστείτε τα αποτελέσματά σα με την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό για μα. και ελπίζω να πάρω μια συγκεκριμένη απάντηση. Να μην μου ξεγλιστρήσετε, να μου δώσετε συγκεκριμένη απάντηση. Αν πράγματι επιβεβαιώνετε ότι είσαστε πρόθυμοι να το κάνετε αυτό. Για ένα λεπτό, κυρία υποψήφια Επίτροπο. Καταρχά, κυρία Στρίκ, να πω ότι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την Τουρκία και με τη Λιβύη δεν είναι αυτή που βλάπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταναστών. Δεν είναι η συνεργασία που τα βλάπτει. Τα δικαιώματα μεταναστών βλάπτονται και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όχι λόγω της συνεργασίας, μέσω της συνεργασίας με τις αρχές μας της Ευρωπαϊκής Ενώσης που να βοηθήσουμε τους μετανάστες. πρέπει να συνεχίσουμε να συνάπτουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Σημαντικό τμήμα αυτού του είδους συμφωνίας θα πρέπει να είναι να δημιουργηθούν νόμιμες διαδρομές τρόποι εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτού του είδους τη συνεργασία με τρίτες χώρες όσον αφορά τη μετανάστευση. Με τα χαράς να ενημερώνω το Κοινοβούλιο και να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις διαβουλεύσεις για αυτού του είδους ε, συμφωνίες. Ευχαριστούμε. Ταρντίνο. Τους... Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Συνδέω την ερώτησή μου αυτή του του συναδέλφου. Δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση. Αναφέρεστε για ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης. Γνωρίζουμε σήμερα ότι όλα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα εντός μεταναστευτικής πολιτικής. Και σήμερα αντικειμενικά χρεοκόπησε η πολιτική και οι χώρε πρώτη υποδοχή έχουν μόνε του μείνει να διαχειριστούν αυτό το πολύ μεγάλο φαινόμενο. Θα καταλάβω ακριβώ τι προτίθεστε, τι εννοείτε όταν μιλάτε για ισορροπημένο συμβιβασμό. Αν μιλάτε για νέα μορφή κατανομή που δεν θα είναι απλώς ε, αλληλέγγυα ή να περιοριστούν ανάντι στην αρχή οι μετασταυτικές ροές. Το μετασταυτικό φαινόμενο θα το διαχειριζόμαστε βάσει ψευτοσυμφωνίας εθελοντικής προσωρινής που έχουν υπογράψει τέσσερις χώρες όπως έγινε πρόσφατα. Τέτοιου είδους συμφωνίες εννοείται. Κυρία Γιωχάνσον, δώστε την απάντηση παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σίγουρη εάν κατανόησα πλήρως το ερώτημά σας, αλλά μπορείτε να υποβάλλετε διευκρινιστική. Τα κρατη μέρη αντιμετωπίζουν διαφορετικές πραγματικότητες και βέβαια έχουμε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και σε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ευρωπαϊκές γεωγραφικές πραγματικότητες. Χαζόμαστε ένα μηχανισμό αλληλεγγύης ούτως ώστε να γίνεται μια σωστή κατανομή των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ρωτήσατε από ό,τι κατάλαβα αν πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέμα σπανάστευση εκτό Ευρωπαϊκή Ενώση. Σωστά. Σωστά, το κατανόησα. Αυτή ήταν η ερώτησή σα. Μπορείτε να διευκρινίσετε, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Ταρντίνου εκτό. Τι, προτι... τι εννοείτε όταν μιλάτε για ισορροπημένο συμβιβασμό. Οι μεταστατικέ ροέ. Στη μεταστευτική πολιτική θα, θα αντιμετωπίζονται Υποχρεωτικά, θα γίνεται κατανομή θελοντικά ή υποχρεωτικά. Θα θέλαμε διευκρινήσει πάνω σε αυτό, όσον αφορά τη διαχείριση των μεταστατικών ροών. Το καταλάβατε τώρα, απαντάει η κυρία Επίτροπο, όπω έλεγε και στον κύριο Μωράη, δύσκολο αυτό να βρούμε κοινό τόπο, βλέποντα ότι έχει αποτελματωθεί κατάσταση στο Συμβούλιο μαζί με τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να έχω όλε τι απαντήσει που ξεκινήσω ε, την προσπάθεια να απεμπλακεί κατάσταση, αλλά να είμαι σαφή για ένα πράγμα. Δηλαδή, ο μηχανισμό αλληλεγγύη δεν είναι εθελοντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε να ισχύει κάτι τέτοιο στου μηχανισμού. Θα πρέπει να βοηθούμε οι μεν του δε στην Ένωση. Συγκεκριμένο τρόπο να γίνει αυτό υπάρχει. Αφού αξιολογήσω την κατάσταση, θα πρέπει να δω ποιο είναι το επόμενο βήμα για το νέο σύμφωνο για το άσυλο και την μετανάστευση. Θέλετε ένα λεπτό συμπληρωματικό, ε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε απάντηση πραγματική. Άλλη μια ερώτηση. Σύντομη. Μιλήσατε για τήρηση της αρχής μη επαναπρόθεσης και της σωστής, της δίκαιας διαδικασίας και επεξεργασίας που είναι κάτι που εφαρμόζουμε. Σε κάθε διαδικασία που γίνεται σωστά ε, ε, επιβαρύνει κυρίως τις χώρες πρώτης υποδοχής μπορεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα η Ευρώπη, δηλαδή το πρόβλημα του κόστου αυτών των διαδικασιών που ακολουθούνται για τις, για Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση, παρακαλώ. Πάλι, αναφέρομαι σε αυτό που απαντήσατε γραπτός. Αναφερθήκατε στην τήρηση της αρχής της μη επιστροφής και της σωστής της δίκαιης διαδικασίας επεξεργασίας των αιτημάτων. Μπορείτε να εγγυηθείτε μια δίκαιη διαδικασία εντός κάθε κράτους μέλους για κάθε μετανάστη. Αυτό είναι κάτι που κοστίζει για κάθε μετανάστη. Πώς προτίθεστε να το καλύψετε. Δηλαδή η Ευρώπη θα επιβαρύνει τα κράτη-μέλη κυρίως αυτά της πρώτης υποδοχής. Αυτές θα υποστούν αυτό το βάρος το οικονομικό. Κυρία Ιωάνντσο. Σας ευχαριστώ. Κάθε χώρα μέλος έχει την υποχρέωση να εξετάσει τις αιτήσει, να τις επεξεργαστεί και να φροντίσει ή να επιστραφούν οι άνθρωποι αυτοί ή αν δεν γίνεται να επιστραφούν λόγω της αρχής του non ρεφουλμαν. τότε αυτό είναι ευθύνη όλων των χωρών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει και να διευκολύνει τι χώρε μέλη να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Αλλά δεν είναι σε θελοντική βάση που ακολουθεί κανεί αυτέ τι θεμελιώδεις αρχέ που εγγράφονται στι συνθήκε μα και βασίζονται και σε διεθνεί ε, συμβάσει. Συνεπώ, η κάθε χώρα μέλο πρέπει να το κάνει. Δεν είναι κάτι που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε, να συνεργαστούμε και γι' αυτό ακριβώς ε, χρειαζόμαστε αυτό το κοινό σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Τώρα ο ε, κύριος Προκατσίνη εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ και καλησπέρα κυρία Γιωχάνσον. Είπατε ότι είσαστε έτοιμοι να στηρίξετε ε, προσωρινά την στήριξη των ανθρώπων αυτών ε, που βρίσκονται στην Μεσόγειο. Υπάρχει εκείνη η δήλωση της Μάλτας που έχουν υπογράψει και άλλοι πριν από 10 μέρες που, σας υπενθυμίζω, μιλάει για πολύ περιορισμένο αριθμό χωρών και θα υλοποιηθεί μόνο για όσους διασώσονται στη θάλασσα. Δεδομένου ότι μόνο το 1% των αφήξεων προέρχονται από τέτοιες δραστηριότητες διάσωσης στη θάλασσα, τι θα κάνετε με τους υπόλοιπους 91% που μας φτάνουν και που μαζικά φτάνουν στις χώρες μας. Πώς θα διασφαλίσετε ότι ό,τι αποφασίστηκε στην Μάλτα δεν θα χρησιμοποιηθεί σαν κίνητρο για να υπάρχουν νέες αφήξεις με τη βοήθεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Απάντηση της κυρίας Γιωχάνσον. Κύριε Ποκασίνη, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας αυτή. Αυτή η προσωρινή συμφωνία της Μάλτας, της Δευτέρας που μας πέρασε, είναι όντως προσωρινή. Θα συζητηθεί, από ό,τι έχω καταλάβει, στο επόμενο Συμβούλιο, την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συμμετέχουν περισσότερες χώρες. Νομίζω ότι αποτελεί ένα βήμα προς τα μπρος. Πρόκειται για μια προσωρινή συμφωνία, αλλά είναι ένα βήμα προς τα μπρος και δείχνει την βούληση των χωρών μελών να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε λύσεις σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Πάντως πρέπει να είμαι και ξεκάθαρη, δηλαδή τέτοιου είδους προσωρινές συμφωνίες δεν αντικαθιστούν μία βιώσιμη λύση για τα ζητήματα ε, της ε, διάσωσης στη θάλασσα. Και δεν συμμερίζομαι την άποψή σα ότι δηλαδή η διάσωση ζών στη θάλασσα, η βοήθεια που τους προσφέρεται να καταλήξουν ε, σε γη, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο. Ένα λεπτό έχετε ακόμα. Δηλαδή τι λέτε, λέτε ότι ε, θα προσπαθήσετε να δουλέψετε προς μια ενιαία προσέγγιση ώστε να μην υπάρχουν προσωρινές λύσεις αν και αυτήν της Μάλτας. Όμως, στα πλαίσια αυτά, μπορείτε δημόσια να δηλώσετε μια για πάντα ότι μόνο αυτοί οι οποίοι πραγματικά διώκονται ή έχουν πόλεμο στις χώρες τους θα φιλοξενούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι οι οικονομικοί ή οι κλιματικοί μετανάστες. Κυρία Κιωχάνσον, απαντήστε παρακαλώ. Κάθε άνθρωπος που κάνει αίτηση για άσυλο έχει το δικαίωμα η αίτησή του να τύχει επεξεργασίας και να καταλήξει σε μία απόφαση για το κατά πόσο δικαιούται κανείς διεθνή προστασία ή όχι. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το ξέρει από πριν, όμως συμφωνώ ότι είναι σημαντικό οι οικονομικοί μετανάστες, για αυτούς πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι, νόμιμοι τρόποι για να φτάνουν στην Ευρώπη ε, για επανεγκατάσταση και να πρόκειται για νόμιμους μετανάστες που φτάνουν στην Ευρώπη για να εργαστούν. Είμαστε μία Ήπειρος που δημογραφικά γυράσκει. Χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο να συνεισφέρει στην οικονομία μας. Εξού και θέλω να βρεθούν νέοι τρόποι και να τους αναπτύξω έτσι ώστε άνθρωποι με προσόντα απ' έξω να έρθουν και να συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Γιωχάνσον. Λιγκουε τώρα. Κορνίλια Χέρντ, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκπλήσωμε που δεν μιλήσατε για τη συνεργασία στον τομέα επιβολή του νόμου. Στι γραπτέ σα απαντήσει, λέτε ότι μία από τις προτεραιότητές σα στον τομέα επιβολή του νόμου είναι να διασφαλίσετε τις απαραίτητες τεχνολογικές καινοτομίες ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε νέες και αναδυόμενες απειλές. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι Εννοείται όταν μιλάτε για τεχνολογικές καινοτομίες. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένο παράδειγμα και πώς θα διασφαλίσετε τέτοιες καινοτομίες ε, να μην παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία τους. Κυρία Γιωχάνσον, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Έρνστ. Είναι πολύ εύστοχη και σημαντική ερώτηση που μου θέσατε. Δύο σημαντικές πτυχές υπάρχουν εδώ. Όταν ε, αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες, βλέπουμε ότι το, το οργανωμένο έγκλημα ε, ε, πολύ γρήγορα τις υιοθετεί και γι' αυτό θα πρέπει να επιταχύνουμε για να μπορούμε να τους καταπολεμήσουμε οι πολίτες μας που πέφτουν θύματα οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας ε, δεν μπορούν να δεχτούν ως απάντηση ότι δεν μπορέσαμε να σας προστατεύσουμε επειδή δεν είχαμε ε, τις νέες τεχνολογίες. Ε, καταλαβαίνω δεν είναι αυτό που λέτε, αλλά είναι σημαντικό αυτό. Όσον αφορά τη χρήση νέων μεθόδων επιβολής του νόμου και προστασίας των πολιτών, είναι σημαντικό ακριβώς να προστατεύουμε τους ανθρώπους ε, και όχι απλά να χρησιμοποιούμε εργαλεία που στόχο έχουν ε, την προστασία των πολιτών. Θα πρέπει να φροντίσουμε να πετυχαίνουμε καλά αποτελέσματα στην πράξη και όχι απλά να προσπαθούμε να δείξουμε τις καλές μας προθέσεις. Θέλουμε αυτά αποτελέσματα για τους πολίτες μας. Πάντα είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μερικές φορές ε, αυτό δεν θεωρείται προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη ήδη από την αρχή όταν αναπτύσσουμε, όταν εκπονούμε νέες προτάσεις στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ, κυρία Έρνστ. Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι τι, πιστεύετε για την χρήση των ε, ε, συστημάτων αναγνώρισης ε, χαρακτηριστικών του προσώπου. Κάτι τέτοιο δεν ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη. Κάποιες χώρες αναπτύσσουν συστήματα παρακολούθησης ολόκληρων πόλεων με βάση την εφαρμογή με βάση εφαρμογέ ε, τη ε, τεχνητή νοημοσύνης, ε, ενώ άλλε χώρε έχουν απαγορεύσει τέτοια χρήση. Εσείς πώς το βλέπετε. Κυρία Έρντ, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν νομίζω ότι θα ήταν σοφό να απαντήσω σήμερα στην ερώτηση αυτή. Θα πρέπει να επανέλθω για να σας δώσω πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Ευχαριστώ κύριε Γιωχάνσον. Περνάμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Θα σας θέσουν ερωτήσεις οι ευρωβουλευτές ε, από τις πολιτικές ομάδες. Χαβιέρ Σασαλέχος, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχετε το λόγο. Κύριε, κυρία Οριστής Επίτροπε, τα τελευταία χρόνια έγιναν διάφορες τρομοκρατικές ε, επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες βέβαια απεφεύχθησαν χάρη στη δράση της αστυνομίας. Σε... Πρόκειται για παντός είδους μορφές τρομοκρατίας που αποτελούν μια πολύ σημαντική απειλή ε, στην ασφάλειά μας. Και ελπίζω την καταπολέμηση της τρομοκρατίας να τη βάλετε πραγματικά ψηλά-ψηλά στους στόχους σας. Σας ερωτώ λοιπόν, Ποια θεωρείτε ότι είναι η κύρια πρόκληση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και τι θα κάνετε. Πιστεύετε ότι η σημερινή αρχιτεκτονική όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία μπορεί να βοηθήσει να αποφευθούν αναδυόμενοι κίνδυνοι. Ή τι θα κάνετε για την επιστροφή ε, τρομοκρατών ή των οικογενειών τους που θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Ε, τι θα κάνετε Επίσης για τα θύματα της τρομοκρατίας σκοπεύετε να υιοθετήσετε μέτρα. Το Κοινοβούλιο είπε ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των θυμάτων από την τρομοκρατία. Απάντηση κύριε Γιωχάντσουρ. Ευχαριστώ κύριε Σαρσελέχος για την ερώτησή σας αυτή όσον αφορά την τρομοκρατία. Είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Ρωτάτε τι είναι το πιο σημαντικό για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Νομίζω ότι είναι η εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε περισσότερη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μελών, μεταξύ αρχών, ε, μεταξύ δυνάμεων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρέπει να χτίσουμε, να αναπτύξουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και βέβαια μπορούμε να βοηθήσουμε και με νέους τρόπους διαλειτουργικότητας, με εμπειρογνώμονες, αλλά το βασικό είναι η εμπιστοσύνη. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα εφόσον συνεργαζόμαστε περισσότερο μεταξύ μας, οι χώρες μέλη δηλαδή και οι αρχές επιβολής του νόμου. Το άλλο είναι η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι ένα καθήκον το οποίο πρέπει να αναλάβουμε ε, συνολικά η κάθε χώρα μέλος με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πραγματογνωμοσύνη σε αυτό το τομέα και είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Τώρα, για τους μαχητές, τρομοκράτες που θέλουν να επιστρέψουν. Αυτή είναι μια απόφαση για την κάθε χώρα μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί όμως να βοηθήσει να διευκολύνει τη συνεργασία έτσι ώστε να διωχτούν, να πάνε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τις τρομοκρατικές τους ενέργειες. Δευτερολογία. Θα ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις για κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για τις απειλές. Στις γραπτές σας απαντήσεις είπατε ότι μόνο έσχατη λύση μπορεί να είναι η επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα, μόνο εφόσον ε, πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς πολύ σημαντικές απειλές. Από την άλλη μεριά, μιλάτε και για τις ε, δευτερογενείς ε, μετακινήσεις που οδήγησαν στην άρση του Σέγγεν σε μερικές περιπτώσεις. Αυτές οι δευτερογενείς μετακινήσεις πιστεύετε ότι απειλούν την ασφάλεια και δικαιολογούν ε, την επαναφορά των συνόρων ε, στα σύνορα μέσα στο χώρο Σέγγεν. Επιπλέον, πιστεύετε ότι μια αναθεώρηση του κώδικα συνόρων ε, του Σέγγεν μπορεί να απαιτείται. Απάντηση, κύριε Γιωχάνσον. Ευχαριστώ. Κύριε Σαρσελέχο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις δευτερογενείς αυτές μετακινήσεις όταν ετοιμάσουμε το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι, αυτό είναι το βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχουμε τρομοκράτες που έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη, δεν μας έρχονται απ' έξω. Έχουν μεγαλώσει εδώ, έχουν ριζασπαστικοποιηθεί εδώ στην Ευρώπη. Οπότε η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί να πετύχει ε, μόνο με ελέγχου στα σύνορα. Σίγουρα όμως ε, πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα για πολλούς και διάφορους λόγους. Το θέμα της τρομοκρατίας όμως είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Ευχαριστώ κύριε Γιωχάνσον. Για σοσιαλιστές, η Μπετίνα Βόλαθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, αναφερθήκατε σε βασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ασφάλεια και συμπροματικές πολιτικές και στόχους σχετικούς. Όμως δυστυχώς αυτό δεν ίσχυσε πάντα. Διαφορετικά νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρούνται παράνομα και κηρύχθηκαν έτσι από το ανώτατο δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Πώ θα εξασφαλίσετε ότι τα μέτρα ασφαλεία θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώ θα εγγυηθείτε ότι οτιδήποτε νέο μέτρο που θεσπίζεται από εσά στον τομέα εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης των συνόρων θα σέβεται αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα περάσει και τη δοκιμασία του δικαστηρίου. Και μία από τις συζητήσεις που λαμβάνει η χώρα όσον αφορά τις δυνατότητες τεχνικές για την επιλογή ε, του νόμου είναι η κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι μια αναγκαιότητα στο σημερινό κόσμο. Συμφωνεί του να επιτρέψουμε τους φορείς τη επιβολή του νόμου να αποκρυπτογραφούν τις επικοινωνίες θα δημιουργήσουν ευάλωτα στοιχεία που θα υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο διαδίκτυο και επικοινωνίες και υπηρεσίε στο διαδίκτυο. Και πώς θα διαφυλάξετε την ε, κρυπτογράφηση των στοιχείων στην Ευρώπη. Κυρία Γιώχανσον, απάντησή σα. Πάντηση Ευχαριστώ κυρία Βόλαθ. Σχετίζεται με πρώτερο ερώτημα αυτό Πρέπει να συνεργαστώ μαζί σας. Όταν θα υποβάλω νέες προτάσεις, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι προετοιμάζονται με τρόπο τέτοιο που θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα εξ αρχής. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε. Στην αρχή πρέπει να τα φροντίσουμε αυτό για την κρυπτογράφηση. όταν διαφαίνονται νέες δυνατότητες να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες εγκληματίες και τρομοκράτες, τότε πρέπει να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε για να καταπολεμήσουμε αυτές τις απειλές. Αυτό είναι κρίσιμο. Όπως προανέφερα όμως, πρέπει να κινηθούμε με έναν τρόπο που θα εξασφαλίζουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ καταπολέμησης της τρομοκρατίας και αύξηση ασφάλειας για τους πολίτες από τη μια και προστασία τη ιδιωτικότητα και θεμελιωδών δικαιωμάτων από την άλλη. Αυτή η ισορροπία πρέπει να είναι σωστή. Για να το πετύχουμε πρέπει να ξέρουμε τι πραγματικά αποτελέσματα επιτυγχάνουμε, τι αντίκτυπο έχουμε για την ασφάλεια. Να μην κάνουμε πράγματα, να μην λάβαμε νέα απόφαση που δεν θα εφαρμόζεται και δεν θα αυξάνει την ασφάλεια για τους πολίτες μας. Αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε όμως ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι που βελτιώνει την ασφάλεια, τότε μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Και πρέπει αυτή την ισορροπία να τη βρούμε μαζί, εσείς και εγώ, και μαζί και με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, κυρία Βόλαθ. Για ένα λεπτό. Αλλάξετε κάτι από αυτό που το Είπατε μετά αξιολόγηση θα μπορούσατε να προβλέψετε μια επικαιροποίηση του κανονισμού Europol, αν αυτό είναι αναγκαίο και εκεί που χρειάζεται. Βλέποντα τα στενά όρια των συνθήκων όσον αφορά την εντολή του Europol, τι είδου επικαιροποίηση προβλέπετε που δεν θα απαιτεί τροποποίηση των συνθήκων, θα δεσμευτείτε ο κανονισμό Europol να συμμορφωθεί με τον κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων για, την, για τα θεσμικά όργανα, φορεί και υπηρεσίες Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ω προβλέπεται από την νομοθεσία. Απάντηση, κυρία Γιωχάνσον. Ευχαριστώ, κυρία Βόλαθ. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσω με τον Επίτροπο, τον Υπεύθυνο για θέματα δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινή ευθύνη μεταξύ, καλύπτεται τα δύο χαρτοφυλάκια μα. με τα χαρά να το συζητήσω αυτό με τον αρμόδιο επίτροπο, τον συνάδελφό μου, θα είναι μόνοι θέματα δικαιοσύνη. Ο κύριος ε, Μάλικ από το ρίνιου Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γιωχάνσον, θα ήθελα να εστιάσω στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, περιμένουν ε, ακόμη μια βιώσιμη πολιτική ασύλου και μετανάστευσης στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι η επιτάχυνση πρωτοβουλειών για ε, ασφαλή καταφύγια για τους ε, πρόσφυγες, για παράδειγμα στη Μόρια, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα είναι αποτελεσματική. Επίσης, η επιτάχυνση των επιστροφών των παράτυπων μεταναστών. Τι θα κάνετε για να γίνει κάτι τέτοιο και τι θα κάνετε για να εφαρμοστεί η οδηγία περί επιστροφής. Και θα αναλάβετε ηγετική θέση μεταξύ των ε, ε, συναδέρφων σας για να αντιμετωπίσετε την παράτυπη μετανάστευση και να καταστρέψετε ε, το κοινικό επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών και να εργαστείτε πάνω σε νόμιμες οδούς. Μπορούν οι πολίτες να περιμένουν από εσά ορατά αποτελέσματα πριν το καλοκαίρι του 2020. Κύριε Γιωχάνσον, μπορείτε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σμάνη. Είναι πράγματι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Ναι, πράγματι θα εντείνω τις προσπάθειες για τις επιστροφές. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, πρέπει να είμαστε πιο σαφείς, πρέπει να έχουμε καλύτερες διαδικασίες και να κλείσουμε τα παραθυράκια. Ε, το κενό δηλαδή που υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς που έχουν δικαίωμα να παραμείνουν και αυτούς που πρέπει να επιστρέψουν. Ε, πρέπει να βελτιωθούμε πολύ στους τομείς αυτούς. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την παράτυπη μετανάστευση και πρέπει να έχουμε στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα αυτών. για να μπορέσουμε να καταστρέψουμε το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών. Αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί που διακινούν ανθρώπους διακινούν και άλλα πράγματα. Διακινούν και πράγματα είναι άνθρωποι που έχουν τεράστιο κέρδος από τις δραστηριότητες αυτές, γι' αυτό πρέπει να καταστρέψουμε το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Πράγματι, θα είναι χρήσιμο να καταλήξουμε σε συμφωνία με τρίτες χώρες και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστώ στενά με τον Αντιπρόεδρο για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής που θα πρέπει να συντονίσει τις προσπάθειες αυτές και θα πρέπει να συνεργαστώ και με τον Επίτροπο για την Γειτονία και τον Αρμόδιο Επίτροπο για ε, τις ε, διεθνείς εταιρικές σχέσεις, νομίζω ότι είναι ο τίτλος του χαρτοφυλακίου. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε λύσεις και νομίζω ότι είναι δυνατόν να βρούμε ε, λύσεις επικεδής και για τις δύο πλευρές αναπτύσσοντας νέες και νόμιμες οδούς μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Όπως σας είπα, ε, έχουμε μεγάλη ανάγκη από ε, εξειδικευμένους εργαζομένους ε, στην Ευρώπη. Επίσης, θέλουμε να αποφύγουμε την διαφυγή των ικανών ανθρώπων. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε καλές συμφωνίες με τρίτες χώρες. κύριε Σμάνι, ένα λεπτό ακόμη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κυρία Γιωχάνσον. Μήπως μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι. Μπορείτε να μας αναφέρετε δύο-τρεις συγκεκριμένες ε, ενέργειες ε, που θα αναλάβετε πριν το καλοκαίρι του 2020, διότι η Ευρώπη θα κριθεί και με βάση ένα συγκεκριμένο θεματολόγιο και ε, συγκεκριμένες πράξεις. Αυτό οφείλουμε στους πολίτες μας και γι' αυτό θα ήθελα από εσά συγκεκριμένες προτάσεις. Κυρία Γιωχάνσον, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, καταλαβαίνω ότι το θέλετε αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι εφόσον εγκρίνεται το διορισμό μου, ε, θα αναλάβω τα καθήκοντά μου. Και η κατάσταση έχει μπλοκάρει εδώ και τρία χρόνια. Η ε, αποστολή μου λοιπόν είναι να ξεμπλοκάρω την κατάσταση, να δημιουργήσω ένα νέο σύμφωνο ασύλου και μετανάστευσης ε, και δεν θα ήταν καθόλου σοφό να ε, σας υποσχεθώ αποτελέσματα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Ελκ, πάλι. Κύριε Βιτσβέγγι, ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα μιλήσω ουγγρικά. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε για τα μέτρα για την αντιμετώπιση της μαζικής μετανάστευσης, εμείς έχουμε αρνητικές εμπειρίες. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά για να κρίνει τις προσπάθειες των ε, χωρών μελών. Υπάρχει η προστασία των εξωτερικών συνόρων που δυστυχώς δεν θεωρείται μέτρο αλληλεγγύης, αντίθετα από ό,τι γίνεται με την υποδοχή μεταναστών. Λοιπόν, πιστεύετε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι ένας τρόπος επίδειξης αλληλεγγύης και τι σκοπεύετε να κάνετε ως επίτροπος για να βάλετε ένα τέλος στα δύο μέτρα και στα δύο σταθμά ώστε κάθε μορφή αλληλεγγύης να μετριέται με τον ίδιο πύχη. Και τι σκοπεύετε να κάνετε ως Επίτροπος προκειμένου τη μαζική αυτή οικονομική μετανάστευση που θέλει να έρθει στην Ευρώπη ή που βρίσκεται εδώ να τυχαίνει διαφορετική αντιμετώπιση από ότι οι πρόσφυγε, οι οποίοι πραγματικά χρειάζονται προστασία. Κύριε Γιωχάνσον, σα ευχαριστώ κύριε Χιντμπέγκη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι μαζικής μετανάστευσης. Το είχαμε το 2015, το 2016, αλλά σήμερα έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο. Όσο ήταν πριν, λίγο πολύ. Ούτε συμφωνώ ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όμως, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι κάτι πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να βοηθάει τις χώρες μέλη να προστατεύουν τα εξωτερικά τους σύνορα. Γι' αυτό και βασιζόμαστε πολύ στην Frontex που πρέπει να μπορέσει να προστατεύσει καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα. Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Frontex είναι ακριβώς αυτό να γίνεται σε συνεργασία με τις χώρες μέλη που πάντα έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τα δικά του σύνορα. Ευχαριστούμε. Ε, λόγο, παρακαλώ, κύριε Μπέγκη. Ευχαριστώ. Κύριε Ρεστίσα, Επίτροπε, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, χώρες προέλευσης, χώρες ε, transit. Τι συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να λάβετε εφόσον οριστείτε ώστε να βοηθήσετε τις χώρες αυτές. Υπάρχει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπει κάλυψη μόνο 5% του κόστους για τέτοιου είδους προγράμματα και δαπάνες. Ενώ οι εμπειρογνώμονε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι έχω καταλάβει, έχουν πει ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 15% για την ίδια περίοδο. Απάντηση, κύριε Ιωάννσον. Ευχαριστώ, κύριε Σβέγγι, για τη συμπληρωματική σας αυτή ερώτηση. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες ε, με τρίτες χώρες διαφέρουν από χώρα σε χώρα και το λέω ήδη ευθύ εξ αρχή ότι αυτό πρέπει να ε, προχωρήσει σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο αλλά και άλλου επιτρόπους. Οπότε θα επανέλθω και θα το συζητήσω αυτό με την Επιτροπή σας σε ένα μετέπειτα στάδιο. Ξανά σοσιαλιστέ, η συνάδελφο Τάνια Φαγιών. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Γιώχανσον. Θα επανέλθω στο Σέγγεν, διότι πιστεύω πραγματικά ότι απειλείται. Κάνατε σαφή διάκριση μεταξύ μεταρρύθμιση κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευση και του σχετικού συστήματο και την εύρυθμη λειτουργία του Σέγγεν για ε, ελεύθερη διακίνηση. Είπατε στην κατ' απάντηση ότι το να επιστρέψουμε σε εύρυθμα λειτουργούσα περιοχή Σέγγεν θα είναι η βασική πτυχή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Δοθέντω το πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση να βρούμε κάποια σοφή μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου, του ευρωπαϊκού, διότι έχει τα χάλια του και ε, έχει τα χάλια του στο Συμβούλιο κατάσταση. Είναι σοφό να διασυνδέσετε τα δύο στοιχεία, δηλαδή τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του κώδικα για τα σύνορα Σέγγεν. Θα προτείνετε μια νέα νομοθεσία συγκεκριμένη που θα αφορά το Σέγγεν στα πλαίσια του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση θα ξανασχεδιάσετε την παρούσα πρόταση που είναι επιτάπητος και έχει διεξαχθεί πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Τότε πόσο χρόνο θα επιτρέπετε στα κράτη-μέλη να παραβιάζουν τους κανόνες. Διότι είναι παράνομα αυτά που συμβαίνουν και απαράδεκτα. Ευχαριστώ κυρία Φαγιόν. Η κυρία Γιωχάνσον. Ευχαριστώ κυρία Φαγιόν. Χαίρομαι που δέχτηκα αυτήν την ερώτηση. Θα ξεκαθαρίσω πέντε πράγματα. Υπάρχει σχέση μεταξύ Σέγγεν και λειτουργούντο συστήματο ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν δημιουργώ τη σχέση, υπάρχει σχέση. Οι παρόντες κανόνες του Δουβλίνου δεν εφαρμόζονται. Αυτό ισχύει σήμερα. Υπάρχει σχέση λοιπόν. Είναι ευκολότερο να επιλύσουμε τα θέματα ε, ταυτόχρονα. Να είμαι ξεκάθαρη, δεν μπορούμε να περιμένουμε να λυθεί το θέμα των εσωτερικών συνόρων στο Σέγγεν αν πρέπει να περιμένουμε επί μακρόν για να λύσουμε άλλα θέματα. Δεν είναι αποδεκτό να υπάρχει μπλοκάρισμα του Σέγγεν λόγω των άλλων θεμάτων. Αν όλα τα θέματα μπορούν να επιληθούν ταυτόχρονα μέσω της νέας όθησης που έχουν λάβει τα θέματα, αυτό είναι καλό, διότι υπάρχουν σχέσεις μεταξύ αυτών. Κάνατε πολύ δύσκολη και σκληρή δουλειά. Τη γνωρίζω για πολλά από αυτά τα θέματα που πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρούσα για το πακέτο ασύλου. Εκτιμώ το έργο σας, πραγματικά. Ε, ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Χρειάζεται όμως να απεμπλακεί κατάσταση στο Συμβούλιο για να γίνει αυτό. Χρειάζεται διμερής διάλογος με τα κράτη-μέλη. Άρα δεν μπορώ να σας δώσω υποσχέσεις σήμερα. Ελπίζω όμως ότι θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατέθεση. Δεν μπορώ να υποσχεθώ. Ευχαριστώ κυρία Γιώχαντσαν. Άλλο ένα λεπτό εσείς κυρία Φαγιών. Παρ' όλα αυτά ελπίζω ότι δεν θα επιτρέψετε αυτές τις παράνομες πρακτικές των οποίων είμαστε μάρτυρες επί πάνω από μια τριετία να κρατήσουν παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Διότι παρόλο που λέτε ότι υποστηρίζετε τα... Δεν θέτεται σαν προτεραιότητα να ξεκινήσετε διαδικασίες επιβαρβάση κατά των κρατών μελών Όμω δεν σεβόσαστε το θεμελιώδη πυλώνα, την ελεύθερη διακίνηση του Σέγγεν. Πότε περιμένετε τη νέα διεύρυνση του Σέγγεν. Θα μπει η Κροατία. Είναι τεχνική πολιτική διαδικασία που ακολουθείτε αν μια χώρα δεν σέβεται το κράτος δικαίου. Κύριε Γιωχάνσον, απάντηση. Πρέπει να επανέλθω αργότερα στην Επιτροπή σας για την επέκταση του χώρου Σέγγεν με τη συμμετοχή νέων μελών. Θα πρέπει να επανέλθω σε αυτό. Οι διαδικασίες επί παραβάση αποτελούν πάντα ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις χρησιμοποιήσει. Δεν είναι σοφό να ξεκινήσουμε τη νέα θητεία σαν νέα επίτροπος έτσι. Εγώ θα προτιμούσα μέσω διαλόγου με τα κράτη-μέλη να ξεκινήσω ανταυτού. Ευχαριστώ κύριε Γιωχάνσον. Ξανά η πράσινη. Ο κύριος Έρικ Μαρκάρτ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Εδώ κάθομαι. Και θα θέσω στα γερμανικά την ερώτησή μου. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι είναι απλό ε, να προκαλούμε φόβο στους ανθρώπους ε, με βάση τη μετανάστευση αναφέρθηκαν μαζικές μεταναστεύσεις εκεί που δεν τις είδαμε και νομίζω ότι ε, πρέπει να είμαστε περήφανοι όταν μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους. Είναι σημαντικό ότι το είπατε αυτό. Είναι επίσης σημαντικό ότι δεν θεωρείτε ότι είναι παράγοντας προσέλκυσης η διάσωση ανθρώπων στη Μεσόγειο. ούτε ότι τα εξωτερικά ε, σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει να γίνουν πιο επικίνδυνα από την Λιβύη για να μην ε, έρχονται οι άνθρωποι από τη Λιβύη εδώ. Μπορούμε όμως να είμαστε περήφανοι για την κατάσταση στη Μεσόγειο και δεν μπορούμε να στηρίξουμε καλύτερα τις ε, ΜΚΟ στη Μεσόγειο. Πώς μπορούμε να τις στηρίξουμε καλύτερα, τι συγκεκριμένο σχέδιο έχετε ώστε να διασφαλίσετε την ε, διάσωση ανθρώπων στη Μεσόγειο ε, και από κρατικά πλοία. Κυρία Ιωάννσον, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρκαρτ. Μέχρι σήμερα πάνω από 900 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο. Είναι μια συνεχιζόμενη καταστροφή. Πρέπει να σταματήσουμε τους ανθρώπους από το να μπαίνουν στα σκάφη αυτά. Πρέπει να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης προς την Ευρώπη και πρέπει να σταματήσουμε τη δραστηριότητα των διακινητών. Παρότι έχουν χαθεί λιγότερες ζωές φέτος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, Παρ' όλα αυτά είναι ε, τρομερή η κατάσταση. Η δική μου προσέγγιση λοιπόν ε, θα είναι να σταματήσουμε τις δραστηριότητες των διακινητών και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βρουν άλλους τρόπους, όχι να μπαίνουν στα σκάφη αυτά. Τούτου λεχθέντος βέβαια. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σύστημα εντοπισμού και διάσωσης. Και αυτό φυσικά παραμένει υποχρέωση και για τα κράτη-μέλη, αλλά και για άλλους, το να σώσουμε ζωές. Όσον αφορά τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ξέρω ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει κατευθυντήρες γραμμές, διευκρινήσεις, ώστε η πραγματική ανθρωπιστική βοήθεια ποτέ να μην ποινικοποιείται. είναι ένα θέμα το οποίο προσλέπω να εξετάσω πιο προσεκτικά και ίσως αυτός να είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάρκαρτ, άλλο ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι ίσως ε, να μην μπορείτε εδώ να μας δώσετε πολύ συγκεκριμένες ε, απαντήσεις, αλλά είναι και δύσκολο για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Λιβύη, όπου ε, γίνεται σε πόλεμος, ε, μπορεί να μην έχουν άλλη επιλογή από το να μπουν ε, στα σκάφια να περάσουν τη Μεσόγειο. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι κάθε μέρα πνίγονται άνθρωποι. Και θα πρέπει ακριβώς να δημιουργηθούν κατευθυντήριες γραμμές ώστε να μην ποινικοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια, ώστε τουλάχιστον η κατάσταση που είχαμε πριν ε, να ε, επικρατήσει, να μην πρέπει να μπαίνουν σε φυλακή οι καπετάνιοι σκαφών που σώζουν ανθρώπους, ε, να σώζουν ανθρώπους και τα σκάφη του Frontex. Μπορείτε να μου πείτε ότι θέλετε να επαναφέρετε την κατάσταση αυτή και μπορείτε να μου πείτε πολύ συγκεκριμένα τι πρόκειται να κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμπληρωματική ερώτηση λοιπόν. Μπορείτε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Μάρκαρτ. Οι πρόσφυγες που είναι αποκλεισμένοι και που ζουν υπό συνθήκες φρικτές, τις οποίες δεν θα έπρεπε να δεχτεί κανένας άνθρωπος, για τους ανθρώπους αυτούς η λύση δεν είναι να μπαίνουν σε επικίνδυνα σκάφη και να προσπαθούν να περάσουν τη Μεσόγειο. Η λύση θα είναι να συνεργαστούμε με άλλους παράγοντες για να δημιουργήσουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να ε, ενισχύσουμε το σύστημα της επανεγκατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το ID. Παρακαλώ. Ο κύριος Κόφοντ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω δανέζικα. Ως Δανός ε, βλέπω μεγάλη ανησυχία την χαοτική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η, ε, η πολιτική ε, μετανάστευση της σουηδικής κυβέρνησης. Βλέπουμε, βλέπουμε να σκάνε βόμβες, βλέπουμε εγκληματικότητα, βλέπουμε πολλά σοβαρά προβλήματα στη Σουηδία και βλέπω ότι ε, εσείς ε, ε, νιώθετε περηφάνεια που έχετε δημιουργήσει την κατάσταση αυτή στη Σουηδία. Είπατε περήφανοι. Ακόμα και οι δανείοι συνάδελφοι από την αριστερά ανησυχούν όσον αφορά την κατάσταση και τις εισόδου ανθρώπων από τη Σουηδία στη Δανία. Έχει ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο και είναι τραγική. Γι' αυτό ερωτώ εάν γίνετε επίτροπος θα προσπαθήσετε να εξάγετε αυτήν την λάθος πολιτική της Σουηδίας στο υπόλοιπο της Σουηδίας και πολύ σωστά ε, θέλετε να εμποδίσετε χώρες όπως τη Δανία να έχουν δικό τους ε, συνοριακό έλεγχο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Κόφοντ. Καταρχά πρέπει να σα πω ότι δεν συμφωνώ μαζί σα όσον αφορά την κατάσταση στη Σουηδία. Επαναλαμβάνω, είμαι περήφανη που η Σουηδία μπόρεσε να προσφέρει καταφύγιο σε τόσο πολλού ανθρώπου κατά τη διάρκεια τη μεταναστευτική κρίση. Αλλά ήδη τότε ήταν σαφές για μένα ότι δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό κοινό σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης. Αυτό είναι σαφές. Ω ε, Σουηδή Επίτροπο δεν θα επιβάλλω Σουηδικέ λύσει, θα είμαι Ευρωπαία Επίτροπο και θα προτείνω ευρωπαϊκέ λύσει, τι οποίε θα αναπτύξω σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το υπόλοιπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Κόφοντ, άλλο ένα λεπτό έχετε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν απαντήσατε ακριβώ στι ερωτήσει μου. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται ε, εφόσον μεγάλη πολιτική πλειοψηφία στο Δανέζικο Κοινοβούλιο ε, πάνε στην Κομισιόν και πούνε ότι θέλουμε να ε, παρατείνουμε τους εθνικούς μας ελέγχους. Και το κάνει αυτό επανειλημμένα, διότι Όλα τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δανών και των πολιτικών του, των εκλεγμένων πολιτικών του, στο ε, ε, Εθνικό μας Κοινοβούλιο, στηρίζουν τον έλεγχο στα εθνικά μας σύνορα. Εσείς λοιπόν ως Επίτροπος θα το παραβλέψετε αυτό και θα πείτε στην πλειοψηφία των δανών πολιτικών ότι δεν επιτρέπεται να το κάνετε αυτό ή θα δεχτείτε ε, το απόλυτα νόμιμο συμφέρον των δανών να μπορούν να ελέγχουν ποιοι εισέρχονται στη χώρα μας. Ε, κυρία Γιωχάνσον, μπορείτε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ήδη θίξει το θέμα αυτό σε προηγούμενες ερωτήσεις. Η εσωτερική εθνική έλεγχη δεν γίνονται ε, σύμφωνα με τους κανόνες του Σέγγεν και γι' αυτό πρέπει να επανέλθουμε σε μια απόλυτα λειτουργική περιοχή Σέγγεν και αυτό είναι απόλυτα ε, σαφές στοιχείο της εντολής μου. Ευχαριστώ το ECR ο κύριος Χόρχε ε, Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ισπανικά θα μιλήσω. Στις απαντήσεις σας, στις γραπτές ερωτήσεις προς την Επιτροπή μας, είπατε ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διάσωση ανθρώπων στη Μεσόγειο και ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτό. Όμως, συγχρόνως, είπατε ότι θέλετε να μπορέσετε να βρείτε τρόπους να αντιμετωπίσετε και να καταρρύψετε τέλος πάντων τον τρόπο δράσης των λαθροδιακινητών. Η κοινή γνώμη στην Ισπανία για παράδειγμα και όχι μόνο διαπιστώνει ότι μερικές φορές συνεργάζονται κάποιες με κυβερνητικέ οργανώσεις με τις διάφορες μαφίες ε, διακινητών. Εσείς ε, τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βρίσκεται μονίμως από την άλλη μεριά σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρνουν οι χώρες μέλη ή όχι. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πισαλπιδάλμπα για την ερώτησή σας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να σεβόμαστε την ανθρωπιστική βοήθεια στη θάλασσα και πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις δρούν προ αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Συνεπώ, δεν θα πρέπει να το μπερδεύουμε αυτό με τους λάθροδιακινητέ. Όπω είπα και νωρίτερα σε απάντηση σε μια άλλη ερώτηση, ε, ζητήθηκαν κατευθυντήριε γραμμέ όταν πρόκειται για συνεργασία με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και ευχαρίστω να το κοιτάξω αυτό μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπονήσουμε τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές. Δεν ξέρω αν έτσι απαντάω στην ερώτησή σας. Ε, δεύτερη ερώτηση. Όχι, νομίζω ότι δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου. Προφανώς η ερώτηση είναι εάν στις περιπτώσεις όπου διοικητικά ή ποινικά διαπιστώνεται από μία χώρα μέλος ότι υπάρχει τέτοια διασύνδεση με κυβερνητικέ οργάνωση με μαφίε όσον αφορά τη διάσωση στη Μεσόγειο, πώ θα τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σεβαστεί την οδηγία διευκόλυνσης που λέει ότι η χώρα μέλος θα αποφασίσει για κυρώσεις ή μέσω δηλώσεων και πρωτοβουλειών πολιτικών παντός είδους θα ε, προσπαθήσει να παρακάμψει αποφάσεις των χωρών μελών ή όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι τελικά η προσπάθεια προστασίας στην Ευρώπη ή η διατήρηση του Σέγγεν θα είναι κάτι που θα υπερισχύσει. Κυρία Γιωχάνσον. Ασφαλώς και οι χώρες μέλη πρέπει να οδηγούν στη δικαιοσύνη τους λαρθοδιακινητές. Εννοείται, αυτό είναι ο ρόλος των αρχών επιβολής ε, του νόμου. Όμως πρέπει συγχρόνως να πω ότι εκείνοι που πραγματικά προβαίνουν σε ανθρωπιστική δράση δεν πρέπει να ποινικοποιούνται. Οι πράξεις τους δηλαδή αυτών δεν πρέπει να ποινικοποιούνται. Ευχαριστώ κύριε Γιωχάνσον. Πάμε στο ΕΛΚ ξανά. Η κυρία Λίνα Ντυπού έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιωχάνσον. Η συζήτηση μέχρι τώρα έδειξε ακριβώς ότι το άσυλο και η μετανάστευση θα αποτελέσει πολύ σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου σας. Ε, αναφέρατε ότι ε, τώρα με τη νέα θητεία, ε, με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπάρξει πάλι κίνηση στα θέματα αυτά. Εγώ ερωτώ, μπορούμε να περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις μέσα στις πρώτες εκατομέρες, για παράδειγμα, και εάν ναι, τι μορφή θα έχουν. Από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλετε να δημιουργήσετε μια τελείως καινούρια ε, δέσμη μέτρων, ε, αλλά εάν ναι, τι μορφή θα έχει και ποια θα είναι η διαδικασία σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιωχάνσον. Ευχαριστώ, κυρία Αντιπό, για αυτή την ερώτηση. δεν θα έχετε συγκεκριμένη απάντηση. Διότι η πρώτη στήμου προτεραιότης είναι να πεμπλακεί κατάσταση. Να βρούμε κοινό έδαφος για ένα νέο σύμφωνο μετανάστευση και άσυλο. Θα είναι δύσκολο αυτό και άλλοι προσπάθησαν πριν από μένα. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε υποσχεθώ ποιε θα είναι οι νέε προτάσει και ποια θα προωθήσω. Ελπίζω να συνεχίσουμε αυτές που έχει εξετάσει και έχει προωθεί στο Κοινοβούλιο. Μπορώ να σας δώσω υποσχέσεις και να δώσω συγκεκριμένη απάντηση. Πρέπει αυτό να αποφασιστεί μετά από διάλογο με τα κράτη-μέλη για να μπορέσει να απευλακεί η κατάσταση. Και δεν νομίζω ότι στις πρώτες 100 ημέρες θα υπάρξουν νέες προτάσεις. Ευχαριστώ. Ακόμα ένα λεπτό έχετε, κύριε ähm, nicht Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένη με την απάντηση αυτή. Θα ε, φτάσω σε άλλο θέμα που θύχτηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Είπατε ότι θέλετε μία νέα βιώσιμη προσέγγιση για τον εντοπισμό και τη διάσωση, search and rescue. Ταυτόχρονα είπατε ότι πρέπει να αποτρέπουμε τους ανθρώπους από το να μπαίνουν ε, στα σκάφη αυτά, αν θέλουμε να σώσουμε τη ζωή τους. Ε, αναφερθήκατε στην καταπολέμηση των δραστηριοτήτων των ε, διακινητών. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα για να ε, καταστρέψετε το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να αποτρέψετε τις εγκληματικές αυτές ενέργειες και πώς θα μπορέσουμε να αποθαρρύνουμε τους ανθρώπους από το να μπαίνουν στα σκάφια αυτά. Ευχαριστώ. Έχετε ξανά το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Τυπού. Συμφωνώ απόλυτα δεν θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μπαίνουν στις βάρκες, καταρχάς. Γι' αυτό θα είναι το σημαντικό να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες, να συνάψουμε συμφωνίες. Ξέρω ότι αυτές οι χώρες δεν θέλουν αυτούς τους διακινητές και τους οργανωμένους εγκληματίες να δρουν στη χώρα τους για να επιβιβάζονται αυτοί οι άνθρωποι στα πλοία, να τους φορτώνουν στα πλοία. Πρέπει να συνεργαστούμε μέσω συμφωνιών με τρίτες χώρες. Πρέπει να εστιαστούμε επί καλύτερων νόμιμων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ρινιού τώρα. Ζαν Κριστόφ Κρετιάν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητή κυρία υποψήφια επίτροπε. Ο κ. Έτιαν, μάλλον. Μας λέτε επανειλημμένα ότι θέλετε να προτείνετε ένα νέο σύμφωνο για άσυλο και μετανάστευση. Θέλετε συμβιβασμό και συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Να σας πω ότι το Κοινοβούλιο από την πλευρά του έκανε αυτό που έπρεπε, τη δουλειά του. Ψηφίσαμε μία εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Στις γραπτές απαντήσεις είπατε ότι θα, θα βασιστούμε στα μέχρι τούδε επιτευθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την νέα προσέγγιση. Το πρόβλημα δεν είναι μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα έγκυται εντός του Συμβουλίου. Θέλω να καταλάβω γιατί θεωρείτε ότι η απόσυρση που αναφέρεται, απόσυρση των προτάσεων για το σύστημα το ευρωπαϊκό το κοινό για το άσυλο, γιατί η απόσυρση αυτών των προτάσεων μπορεί να οδηγήσει σε απεμπλοκή των εργασιών του Συμβουλίου. Γιατί θεωρείτε ότι μια τέτοια κίνηση θα διτουργήσει Απάντηση κύριε Γιώχανσον. Ευχαριστώ κύριε Τιέν. Είναι εύλογη ερώτηση και καταλαβαίνετε ότι έχω δυσκολίες και δεν μπορώ να δώσω όπως αναμένεται συγκεκριμένη απάντηση για αυτά τα θέματα. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση. Αυτή η αποτελμάτωση στο Συμβούλιο πρέπει να λυθεί, να σταματήσει. Η αποστολή από την εκλεγήσα πρόεδρο, πρόεδρο είναι να έχουμε ευρύτερη προσέγγιση από το πακέτο το άσυλο, να βρούμε λύση και για τη μετανάστευση και για το άσυλο. Αυτό αποτελεί προτεραιότητά μου. Να αναπτύξω το νέο σύμφωνο αυτό. Για να το κάνω αυτό, κάποιοι θεωρούν ότι είναι σαν τι επικίνδυνες αποστολέ. Να βρούμε κοινό τόπο στο Συμβούλιο. Δεν πιστεύω. Νομίζω ότι γίνεται. Πρέπει να είμαι όμως πολύ προσεκτική. Να μην δέσω τα χέρια μου και να μην μπορώ να κινηθώ μετά. Πρέπει να ελέγξω τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να αποσύρουμε κάποιες προτάσεις και που έχουν προωθηθεί σαν μέτρα στο Κοινοβούλιο. Αλλά δεν μπορώ απ' την άλλη να υποσχεθώ ότι δεν θα το κάνουμε αυτό. Αυτή είναι η απάντηση. Ξανά εσείς, κύριε Τιέν. Ευχαριστώ κυρία Γιώχανσον. Το Κοινοβούλιο θα ήθελε να έχουμε ένα επίτευγμα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και καταλαβαίνω γιατί θέλετε να διαβρύνετε το πλαίσιο και να λάβετε υπόψη και τα θέματα μετανάστευσης. Θέλετε να λάβετε υπόψη και θέματα των συνόρων, του ελέγχου των συνόρων και τα θέματα του Σέγγεν ή πιστεύετε ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να είναι εκτός των θεμάτων ασύλου και μετανάστευση. ή θέλετε να τα εντάξετε μέσα σε ένα πακέτο και αυτά. Η απάντησή σας κύριε Γιωχάνσον πρέπει να επανέλθω στο περιεχόμενο του νέου συμφώνου, που το επανεξετάσω ότι πρέπει να είναι στο νέο σύμφωνο. Πολλά είναι επιτάπητο ταυτόχρονα. Και από την εμπειρία μου, καμιά φορά, όταν ισχύει αυτό, είναι να απεμπλέκεις μπλοκαρισμένες καταστάσεις Τώρα, κατά πόσο όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν, αυτά που αναφέρατε σε ένα πακέτο, επανέλθω αργότερα. Τώρα, περνάμε στους μη εγγεγραμμένους. Ο κύριος Φεράρα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Η κυρία Φεράρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά, υποψήφια επίτροπε, για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση ελπίζω να μην οδηγήσει σε απόσυρση των χαρτοφυλακίων που έχουν αποτελματωθεί στο Συμβούλιο. Διότι μάλιστα ω εισηγήτρια του κανονισμού για τη διδικασία σύλλου μπορώ να είμαι μάρτυρε των τεράστιων προσπαθειών που έκανε το Κοινοβούλιο για να καταλήξει μια λύση που θα μπορούσε να είναι βιώσιμη παντού οριζόντια και να μπορέσει να προσφραστεί την ε, προσέγγιση σε πακέτο για να μην υπάρχουν ασορροπίες μεταξύ των κρατών μελών και να μην υπάρχει μεταστευτική πολιτική που θα είναι αναποτελεσματική όσον αφορά το νέο πακέτο. Πιστεύετε ότι μπορεί να αποτελέσει τμήμα αυτού. Η νόμιμη διαδρομή για να μπει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμιμες λύσεις. Θα δώσετε συνέχεια στην έκθεση Λόπε Αγγιγιάρ για τις ανθρωπιστικές θεωρήσει και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχή σε τρίτε χώρε στη Νότια Μεσόγειο, ούτως ώστε να μπορούν εκεί να ζητήσουν προστασία ανθρωπιστικοί οι άνθρωποι στην νότια ακτή του Μεσογείου, αντί να πρέπει να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Ίσως ε, θα μπορούν να διχειρίζονται αυτά τα κέντρα, να τα διχειρίζεται η Πατιαμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Η απάντησή σας, κυρία Γιωχάνσον. Σας ευχαριστώ, κυρία Φεράρα. Όπως είπα και στην αρχική μου παρουσίαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και εσείς προσωπικά έχετε κάνει πολλή δουλειά πάνω στους φακέλους αυτούς. Έχετε πετύχει συμβασμούς, καλή συνεργασία και το εκτιμάω όλος ιδιαίτερος. Αυτό είναι ένας πραγματικά ευρωπαϊκός τρόπος συνεργασίας, να πετυχαίνουμε συμβιβασμούς, γεφυρώνοντας τις διαφορές μας, ε, τις πολιτικές και άλλες. Και αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Συγχρόνως, η απόσυρση μιας τέτοιας πρότασης δεν αποτελεί λύση. Πρέπει όμως να βρω τρόπο να προχωρήσουμε και γι' αυτό δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Αλλά ναι, νόμιμη οδή. Αυτό πρέπει να αποτελέσει μέρος του νέου συμφώνου, η δημιουργία δηλαδή τέτοιων νόμιμων οδών. Πρέπει να είναι μέρος του νέου συμφώνου μετανάστευσης και ασύλου, ναι και γνωρίζω την πρόταση για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Θα μπορούσε να συζητηθεί, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτό, αλλά συγχρόνως πρέπει να πω ότι είναι κάπως εύκολο να μιλάμε για επανεγκατάσταση και ανθρωπιστικούς διαδρόμους που έχουν ήδη λειτουργήσει καλά κατά το παρελθόν. Έτσι καλώς όμως η συζήτηση θα συνεχιστεί για αυτά τα θέματα. Έχετε ένα λεπτό ακόμα κύριε Φερέρα. Ευχαριστώ. Να πάω σε άλλο πεδίο, τη εσωτερική ασφάλεια, κυρίω όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε προτεραιότητα ή πρόθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσετε συνέχεια στην έκθεση ΚΡΙΜ. Δηλαδή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρξει νομοθεσία για να καταπολεθεί το οργανωμένο έγκλημα, όπω και τα οργανώσει τύπου Μαφία. Είναι ένα διεθνέ φαινόμενο και αποθαρρύνεται και εμπιστοσύνη των ε, πολιτών εναντί των δημοσίων θεσμών τα παραβίαση των ανθρώπινων δικαιώματα. Όσον αφορά την οδηγία για το child sexual abuse και το child exploitation, τι προτίθεστε να κάνετε για να εγγυηθείτε ότι τα κράτη-μέλη θα συμμορφωθούν απόλυτα και τι δράσεις θα νομολογήσετε για την εντεντικοποίηση της, κατάστασης της ε, σεξουαλικής ε, κακομεταχείρισης των ανηλίκων, ειδικά προγράμματα για εκείνους που παραβιάζουν τις, ε, την νομοθεσία και πώς θα υποστηρίξετε και τα θύματα μετά. Απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. πράγματι είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά. Το οργανωμένο έγκλημα και οι μαφιόζικες οργανώσεις αποτελούν δηλητήριο για τις κοινωνίες μας. Χρειάζεται συνοχή στην κοινωνία και το αντίθετο συμβαίνει με αυτέ. Δεν πρόκειται μόνο για τα θύματα δηλαδή των εγκληματικών αυτών ενεργειών, πρόκειται για ολόκληρη την κοινωνία η οποία υποφέρει. Γι' αυτό και πρέπει να σταματήσει αυτό το δηλητήριο. Τώρα πρέπει να επανέλθω όσον αφορά τι συγκεκριμένε δράσει όταν αναλάβω τα καθήκοντά μου. Τότε μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένα για τα βήματα που πρέπει να αναλάβουμε. Ξέρω όμω ότι υπάρχουν πολλέ προτάσει που έχουν ήδη υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε πάρα πολύ στην υλοποίηση, την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. Μην αποκλείεται όμως ότι, το ότι θα συνεχίσουμε και με άλλες προτάσεις ε, στο ίδιο θέμα, αλλά θα επανέλθω από αυτού. Το ίδιο ισχύει και ε, για το θέμα της κακοποίησης των παιδιών σεξουαλικής κακοποίησης. Η πορνογραφία, για παράδειγμα, μα το κέντρο της βρίσκεται στην Ευρώπη, μην το ξεχνάμε, στις χώρες μέλη. Είναι ένα τρομερό έγκλημα αυτό. Και πρέπει και εδώ να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών επιβολής του νόμου για να πάψουμε να έχουμε αυτό το κλιματικό φαινόμενο της πορνογραφίας και της ε, σεξουαλικής κακοποίησης. Συνεχίζουμε. ECD και από εδώ είναι επόμενος ο μιλητής μας, ο Πιέτρο Μπαρτόλο, που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Τους μετανάστευσης. Καλησπέρα. Δεν ακούγεται δυστυχώ ο μιλητή. Α, ναι, Επιστολή σα, Είπατε ότι θέλετε να εξεργαστείτε νέα προϊόσιμη προσέγγιση, αξιόπιστη προσέγγιση όσον αφορά την έρευνα και διάσωση. Στη γραπτή σα απάντηση είπατε ότι η εμπειρία των τελευταίων μηνών έθεσε στο φω το βασικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη και τον συντονισμό των δράσεων για τη μετεγκατάσταση και την κατανομή των ατόμων που είναι στα πλοία μετά την αποβίβαση στα κράτη-μέλη. Η έρευνα και διάσωση ρυθμίζεται από τη Διεθνή Νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταρχήν αρμοδιότητες συντονισμού. Αληθεύει όμω ότι μπορεί να κάνει περισσότερα δίνοντα υποστήριξη οικονομική και ηλική στα κράτη-μέλη για την ενίσχυση τη δυνατότητα που έχουν να διασώσουν ζωέ στη θάλασσα. Τι δράση συγκεκριμένα, τι πρωτοβουλία θα υθετήσετε για να συμμορφωθείτε με την υποχρέωση που, που έχετε γράψει στην επιστολή σα, δηλαδή να υπάρχει αξιόπιστη προσέγγιση και μόνιμη για την έρευνα και διάσωση. Ακούσα την ερώτηση, κυρία Γιώχανσον, απαντήστε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βαρτόλο, είπατε, όντως έχει ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει εδώ. Και τώρα έχει παίξει αυτό το ρόλο συντονισμού δηλαδή και διευκόλυνσης προκειμένου να βοηθήσουμε ολόκληρη την αλυσίδα όταν έχουμε να κάνουμε τον εντοπισμό και τη διάσωση γιατί πρόκειται και για το πώς θα φτάσουν ε, στην χώρα, όποια χώρα είναι αυτή, ε, όλη τη διαδικασία για αίτηση ασύλου δεχομένως και τα λοιπά. Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη αλυσίδα εδώ που θα αποτελέσει μέρος ε, της συνολικής λύσης που μου ζήτησε να εκπονήσω η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Μπαρτόλη για ένα λεπτό ακόμα. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιο συγκεκριμένα, βάσει τις απαντήσεις που έχετε δώσει, ποια είναι τα σχέδιά σα και επιλογέ σα για να μετωπιστεί το θέμα τη έρευνα και διάσωση βάσει τη αρχή τη αλληλεγγύη. Σύμφωνα με την αλληλεγγύη, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μοιραστούν εξίσου την ευθύνη των ετούντων άσυλο σε πλήρη σεβασμό των αρχών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και θεμελιωδών δικαιωμάτων και του Διεθνού δικαίου. Παρακαλώ, η οριστής Επίτροπος να απαντήσει. Ευχαριστώ. Πρόσφατα είχαμε μια προκαταρτική συμφωνία της ε, Μάλτας για τέσσερις χώρες και είναι κάτι που φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί στο Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Οπότε θα δούμε τι θα βγει από αυτές τις συζητήσεις. Εγώ έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα άνοιγμα και μια επικοδομητική προσέγγιση από τις χώρες μέλη. Ελπίζω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Οπότε επιτρέψτε μου να επανέλθω στον διάλογό μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια μετέπειτα στιγμή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. ΕΛΚ. Η κυρία Ναντίν Μορανό τώρα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γαλλικά, Πρόεδρε. Κύριε Οριστή, Επίτροπε, με εκπλήσει πως τις γραπτές σας απαντήσεις για την καταπολέμηση της παράτυπης, παράνομης μετανάστευσης, το μόνο που λέτε είναι να βρεθούν νόμιμοι οδοί για την νόμιμη μετανάστευση. Δεν μιλάτε για το πώς θα επιστρέψουν οι παράνομοι στις χώρες τους, ώστε το μεταναστευτικό να το αντιμετωπίζουμε με τρόπο απόλυτο, ανθρωπιστικό μεν, αλλά απόλυτο. Εντάξει, μιλάμε για τα δικαιώματά τους, αλλά όταν έχουμε αποφάσεις της δικαιοσύνης για την επαναπρόθεση των ανθρώπων αυτών, αυτές δεν τηρούνται, δεν υλοποιούνται, οπότε το μόνο που λέμε είναι δικαιώματα για το άσυλο. Ενώ το αποφασίζεται από διάφορες χώρες να φεύγουν και να επιστρέφουν στις χώρες τους, μόνο το 1 τρίτο από αυτού έχει όντω επιστρέψει, ενώ η δικαιοσύνη παίρνει αποφάσει. Τι θα κάνετε λοιπόν για να αυξηθεί δραστικά ο αριθμό των ατόμων που επιστρέφουν, που βρίσκονται δηλαδή παράτυπα στι χώρε μα. Ευχαριστώ, κύριε Μωρανό. Όντω είναι μια πολύ σημαντική πτυχή και αυτή. Ε, φυσικά και πρέπει μαζί να φροντίσουμε να αυξηθούν οι επιστροφές των ατόμων που δεν έχουν το δικαίωμα να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως, όπως είπα και στην αρχική μου παρουσίαση, ισχύει. Υπάρχει το δικαίωμα αίτησης ασύλου, υπάρχει το δικαίωμα σε διεθνή προστασία, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιοι έχουν αυτά τα δικαιώματα. Αυτοί που δεν τα έχουν πρέπει να επιστρέφουν. Μέχρι τώρα αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί καλά. Πράγματι το ένα τρίτο μόνο για όσους έχει ληφθεί η απόφαση επιστροφής έχουν πράγματι επιστρέψει. Συνεπώς εδώ πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Όμω δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη η οποία επιστρέφει τον κόσμο. Είναι ευθύνη των χωρών μελών να φροντίσουν για την επανεστηρική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει. Έχουμε συμφωνίε επανεισδοχή με τρίτες χώρες. Ε, μπορούμε να φροντίσουμε για διευκολύνσεις αλλά μπορούμε να συζητήσουμε τι παραπάνω θα μπορούσε ενδεχομένω να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επανεισδοχή αυτή, ώστε να ε, έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει και οι διαδικασίες ε, περί να επιταχυνθούν και αυτό θα βοηθούσε. Ευχαριστούμε. Κυρία Μωρανό, έχετε ένα λεπτό ακόμα. Εγώ περίμενα να μου μιλήσετε για τις συμφωνίες επανεισδοχής. Έχουμε 17 Καμερούν, Μαλή, την Ισία κτλ. Και στην Αφρικανική Ένωση, όπου έχουμε πολλούς που είναι transit, δεν καλύπτονται από τέτοιες συμφωνίες. Είναι μια προτεραιότητα, συμφωνείτε, Έπειτα δίνουμε 17 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη της Αφρικής. Εγώ δεν σας άκουσα ποτέ να μιλάτε για την ευθύνη της Αφρικανικής Ένωσης και των χωρών προέλευσης. Περιμένω την απάντησή σας από αυτού. Εσείς, κυρία Ιωάννησον. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μωράνο. Πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερες συμφωνίες επανεισδοχής με διάφορες χώρες. Όντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει σε αυτό και γνωρίζω ότι σε μερικές περιπτώσεις οι χώρες μέλη έχουν τις δικές τους συμφωνίες. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και τις χώρες μέλη, ώστε να έχουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό σύστημα επανεισδοκής, γιατί είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Η πάλι. Τώρα το λόγο έχει η συνάδελφος, η κυρία Μαλίν Μπιόρκ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Ε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Όπως ακούσατε σήμερα, κάποιοι θέλουν να, επιλέξουμε, να επιλέξει η Ευρώπη τον ίδιο τρόπο με τον Τραμπ, ε, την εκδοχή Ορμπάν, με τύχη και ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλοι από εμά όμως θέλουν άλλα μέτρα. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μία ήπειρος όπου οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν και να θέλουν να έρθουν. Ε, θέλουμε να υπερασπιστούμε την σύμβαση της Γενέβης και θα πρέπει να σταματήσουμε την πολιτική των κλειστών συνόρων. Υπάρχουν ρατσιστές που θέλουν το ε, αυστραλέζικο μοντέλο. Ε, να, χειριζόμαστε, ναι, να διεκπαιρεώνουμε δηλαδή τις αιτήσει ασύλου εκτός ε, της Ευρώπης. Εσύ θα διασφαλίσεις το δικαίωμα αίτησης ασύλου στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω και μια ερώτηση για τη Λιβύη που θα θέσω μετά την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή, κυρία Πιόρκ. Θα απαντήσω όμως στα αγγλικά. Συμφωνώ ότι σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε να απειλείται το δικαίωμα ε, ε, αίτηση ασύλου των ε, μεταναστών. Και αυτό είναι τρομακτικό. Και ακριβώς γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, διότι ο ευρωπαϊκός τρόπος είναι όπως λέει η σύμβασή μας, ε, να υπάρχει το δικαίωμα αίτησης ασύλου. Αυτό αναφέρεται σαφώς στη συνθήκη μας. Ω επίτροπο, λοιπόν θα υπερασπίζομαι πάντα και τις θεμελιώδει αξίες μα και την συνθήκη και είναι απόλυτα σαφέ αυτό και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα μέρη του κόσμου. Το ότι θεσπίζονται σαφώ τα δικαιώματα των μεταναστών να ζητήσουν άσυλο. Έχουμε αυτέ τι σαφεί αξίε τι οποίε υπερασπιζόμαστε. Πολύ ευχαριστώ σε λοιπόν. Θα υπερασπιστώ, ε, θα αγωνιστώ για τα δικαιώματα αυτά και εδώ εντό ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ κυρία Πιόρκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πιο σαφή απάντηση θα απορρίψει προτάσεις για εξοεδαφική διεκπαιρέωση των αιτήσεων. Και η άλλη με ερώτηση ε, ε, έχει να κάνει με την Λιβύη. Είδαμε εδώ παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και διαπιστώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνένοχη. Θα, θα δώσει σε τέλος λοιπόν στην συνεργασία μας με την ακτοφυλακή εκεί. Επίσης είμαι εισηγητής του Κοινοβουλίου για την επανεγκατάσταση. Μπορείς λοιπόν να διασφαλίσεις ε, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ε- Ένωσης ε, για την επανεκατάσταση να βασίζεται στις αρχές του UNHCR και να παραμείνει ανθρωπιστικό. Κυρία Γιωχάνσον, μπορείτε να απαντήσετε. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πιόρκ. Όσον αφορά την Λιβύη, δεν βλέπω πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση στη Λιβύη αν σταματήσει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι οι ακτοφύλακες της Λιβύης παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει την ακτοφυλακή της Λιβύης σε διάφορες πτυχές ε, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις ενέργειές τους. Θα επανέλθουμε στο τι πρέπει να γίνει στη Λιβύη. Πρέπει να πω όμως ότι δεν νομίζω ότι η πάυση της συνεργασίας που έχουμε με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ε, με τον UNHCR, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και η κατάρτιση ε, της ακτοφυλακή της Λιβύης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν βλέπω πώ το τέλος τη συνεργασία αυτή θα βελτιώσει την πολύ δύσκολη, την φρικτή κατάσταση στη Λιβύη. Όσον αφορά την επανεγκατάσταση, η συνεργασία με ε, την ύπατη αρμοστία είναι φυσικά ε, ο ακρογωνιαίος λήθος της εργασίας μας πάνω στην επανεγκατάσταση. Δεν θα απορρίψω όμως σε καμία άλλη πτυχή. Νομίζω ότι η επανεγκατάσταση είναι πολύ σημαντική πτυχή των νομίμων οδών ε, μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσω ε, να ε, το καταφέρω αυτό σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριε Γιωχάνσον από το S&D, ο συνάδελφος Χαβιέρ Μορένο. Παρακαλώ ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Γιωχάνσον πλησιάζουμε στο τέλο. Όπω γνωρίζετε πολύ καλά, η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η προστασία των γυναικών είναι κάτι που βρίσκεται στο κέντρο της δράσης της πολιτικής μας ομάδας. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι θετική δέσμευση που λαμβάνεται όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες μας τις πολιτικές. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω όσον αφορά την καταπολέμηση της λαθροδιακίνησης και την προστασία των θυμάτων, κυρίως των γυναικών και των παιδιών, κυρίως των κοριτσιών. Δυστυχώς, η λαρθιοδεκίνηση οδηγεί σε πολλά θύματα και βέβαια τεράστια κέρδη. Εκατομμύρια κάθε χρόνο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να καταλήξει σε κάποια λύση συνεργασία με τις χώρες μέλη και συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να προστατεύονται τα θύματα και οι υπεύθυνοι να διώκονται από τη δικαιοσύνη. Πώς θα εφαρμόσετε καλά την οδηγία του 2011 για τη λαθροδιακίνηση και για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών και τι μέτρα και με τι οικονομικούς πόρους θα λειτουργήσετε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γιωάννησον, να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μωράνο Μωρένο Σάντσες. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας του 2011, Πρέπει να επανέλθω με συγκεκριμένες δράσεις αργότερα. Αλλά αυτό που πρέπει να πω για την κίνηση είναι κάτι το οποίο με απασχολεί πολύ και ξέρουμε ότι τα μισά εκ των θυμάτων είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόβλημα ε, που έχει να κάνει μόνο με έξω από τα σύνορά μας, όχι, το έχουμε εδώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα περισσότερα θύματα της εμπορίας ε, ανθρώπων έχει θύματα γυναίκες. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχυθεί ο αγώνας μας κατά της εμπορίας ανθρώπων. Και είμαστε έτοιμοι να ε, ψάξουμε να βρούμε νέες νομοθετικές προτάσεις σε αυτό το τομέα. Διότι οι εγκληματίες όντως βγάζουν πάρα πολλά λεφτά χρησιμοποιώντας ε, τα θύματα τους, τα κορίτσια αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω να βρω νέες ε, νομοθετικές προτάσεις, να τις εκπονήσω και να σας τις προτείνω και να δούμε μήπως πρέπει να έχουμε και μια νέα στρατηγική καταπολέμωσης καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει, γιατί είναι τροπή τα μισά από αυτά τα θύματα να είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστούμε κύριε Γιουχάνσον. Ο κύριος Μορένο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Βέβαια δεν είσαστε μόνοι σας στον αγώνα αυτό. Έχετε και τη συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορία ανθρώπων. Έχετε τη Europol και έχετε και το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της εμπορίας ανθρώπων. Πώς θα ενισχύσετε τις εξουσίες όλων αυτών τον τρόπο δράσης τους, πώς θα συνεργαστείτε μαζί τους. Και μια μικρή ερώτηση, υπάρχει ε, ένα, μια κατηγορία που είναι η ανήλικοι, κυρίως η ασυνόδευτοι. Τι θα κάνετε προκειμένου η κατηγορία αυτή που εκτίθεται ε, πάρα πολύ σε κινδύνους είτε για εμπορία ανθρώπων, είτε για εμπορία οργάνων, είτε για σωματεμπορία. Τι θα κάνετε και πώς θα βοηθήσετε τα θύματα αυτά που βρίσκονται στις χώρες μας. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ κύριε Ιωάννησον. Ευχαριστώ κύριε Μωρένο Σάντσεθ. Όλοι αυτοί οι τομεί είναι τομεί για τους οποίους πρέπει να κάνουμε περισσότερα όλοι μαζί. Βέβαια και είμαι υπεύθυνη για ε, πολλά, πολλούς από αυτούς τους οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν. Κυρίως πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την οτροπία της ατιμορρησίας και μετά να βοηθήσουμε τα θύματα. Θα επανέλθω σε εσά αργότερα με προτάσεις μου. Και κυρίως με την αξιολόγηση του κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε νέες προτάσεις ή όχι. Η πράσινη τώρα. Ο κύριος Νταμιέν Καρέμ. Παρακαλώ κύριε Καρέμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γιώχαντσον, ήρθα ε, θετική άποψη όταν ήθελα να ακούσω την ακροασή σας. Κάποια από αυτά που είπατε με ανακούφισαν, ε, ε, πάντως κάποια με ανησυχούν η αριστολογία. Λυσμονείται σε αυτή την άκρωση ότι πίσω από αυτά τα λόγια υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν άντρες, υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν πάρα πολύ και πάρα πολύ νεκροί. Θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε καταπήγουσες απαντήσεις. Καταλάβαμε ότι θέλετε να αποφύγετε να, αυξάνουν, να ανεβαίνουν στο πλοίο αυτοί που ψάχνουν για ε, ε, να είναι πρόσφυγες. Θα πρέπει όμω να ξεκινήσουμε και διάσωση στη θάλασσα για αυτού. Καταλάβαμε ότι θέλετε να απεμπλακούν οι συζητήσει για το Δουβλίνο. Αυτό που είναι κάτι απαραίτητο και ήρθε ο χρόνο ε, να σταματήσουν τα παιχνίδια πάνω σε αυτό. Για τη μέθοδο του Συμβουλίου που μπλοκάρει το θέμα δεν δώσατε απάντηση ψάχνοντα όχι με ειδική πλειοψηφία αλλά με ομοφωνή απάντηση και θέλετε να γίνονται σεβαστέ συνθήκε. και θα πρέπει να πετήσετε από το, από το Συμβούλιο ε, τελικά να αλλάξει και να λάβει αποφάσει με ειδική πλειοψηφία παρά με συνένεση που τελικά είναι μια δικαιολογία για έλλειψη δράση. Και τώρα έχετε την, το χρόνο να απαντήσετε κυρία Γιώχανσον στην ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Καρέμ. Απάντησα πολλές ερωτήσεις για έρευνα και διάσωση. Δεν έχω άλλη απάντηση παρά αυτές που έδωσα. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, έχουμε μια νέα επικοδομητική προσέγγιση. Με αυτή την αρχική συμφωνία στη Μάλτα την περασμένη εβδομάδα θα διεξαχθεί συζήτηση στο αρμόδιο συμβούλιο στο, την επόμενη εβδομάδα, το Συμβούλιο Υπουργών. Ελπίζουμε στο Συμβούλιο Εσωτερικών να βρεθεί μια λύση. Δική μου αποστολή είναι να προτείνω και πιο βιώσιμη προσέγγιση για όλα αυτά. Και πρέπει να επανέλθω στην αξιότιμη επιτροπή σα ε, όσον αφορά το θέμα ε, για την έρευνα και διάσωση στο μέλλον. Όσον αφορά το Δουβλίνο και τον κανονισμό του Δουβλίνου και το χαρτοφυλάκιο που έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, κανένα δεν θα είναι πιο ευχαριστημένο από μένα αν σταματήσει αυτό το μπλοκάρισμα. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, δυστυχώ. Διότι ήδη έχει σημειωθεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι ένα κομμάτι του δυσχερέστατου έργου που με περιμένει, να βρω έναν τρόπο να σταματήσει αυτή η αποτελμάτωση στο Συμβουλίο. Όπως προανέφερα, θα πρέπει ίσως να χρειαστώ όλη μου την εμπειρία και πιθανότατα και κάποιες άλλες προτάσεις επιτάπητος ταυτόχρονα, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκαριστεί η κατάσταση. Προηγουμένως είχα πει σε απάντηση ότι βεβαίως σαν επερχόμενη επίτροπος, εάν με εγκρίνετε, θα ξεκινήσω με ένα διάλογο για να πετύχω την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Στο τέλος όμως πρέπει να λάβουμε απόφαση για ένα νέο σύμφωνο. Ευχαριστώ κυρία Γιώχανσον. Κύριε Καρέμ, η αντίδρασή σας για ένα λεπτό και διευκρινιστική ερώτηση θα πρέπει να αξιολογήσουμε για την εφαρμογή των παρόντων μέτρων πριν ξεκινήσει αυτό το σύμφωνο. Δεσμεύεστε να αξιολογήσετε την εφαρμογή των διαφόρων παρόντων μέσων του πακέτου άσυλο και αν ναι, σε ποια προθεσμία, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το χρονικό διάστημα. Επίση, να φροντίσετε ούτω ώστε κάθε νέα πρόταση θα πρέπει να εδράζεται επί των συμπερασμάτων αυτή τη εκθέσεω για εφαρμογή των μέτρων και να γίνει και μια μελέτη αντικτύπου σε συνεργασία με του εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών. Έχετε το λόγο, κυρία Γιώχανσον. Ήδη έχουμε 7 χαρτοφυλάκια επιτάπητος στο πακέτο ασύλου. Δεν θέλω να ξεκινήσω από το μηδέν. Ελπίζω να μπορέσουμε να βασιστούμε στα επιτευθέντα στο Κοινοβούλιο. Η πρώτη προσέγγιση δεν θα είναι να ξεκινήσω από την αρχή, αλλά να συνεχίσω στα υπάρχοντα. Πρέπει όμως να περάσω αυτή τη διαδικασία, να δω τι χρειάζεται για να πεμπλακεί η κατάσταση. Με τα χαράς να ενημερώνω την Επιτροπή σας για το θέμα και να συνεχίσουμε και τη συνεργασία σε αυτού τους τομείς. Σας ευχαριστούμε. Στο δεύτερο γύρο, τώρα περνάμε στην τελευταία ευθεία. Ο κύριος Πάολο Ραντζέλ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη διορθώνει ο Πρόεδρο. Συγγνώμη, έκανα ένα λάθο. Ναι. Είναι και η ομάδα Renew. Συγγνώμη. όντω, έκανα λάθο. Πρώτη τελευταία ερώτηση από την ομάδα Renew. Μόριτ Κέρνερ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, θα μιλήσω γερμανικά. Κυρία Γιωχάνσον, στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας κάτι πάει στραβά από τις 22 Ισλαμιστικές επιθέσεις από το 2009. Και τουλάχιστον ένας από αυτούς ε, ήταν ήδη γνωστή στην αστυνομία, αλλά και η αστυνομική ε, συνεργασία στην Ευρώπη έπρεπε να βελτιωθεί. Αντί για αυτό όμως απλά συλλέξαμε περισσότερα δεδομένα. Νομίζω ότι θεώρησε κανεί ότι θα είναι πιο εύκολο να βρούμε την ε, βελόνα στα άχυρα αν αυξήσουμε τα άχυρα. Ε, εσείς θα αλλάξετε αυτήν τη λάθος πολιτική ή απλά θα συνεχίσετε τη συλλογή όλο και περισσότερων δεδομένων. Θα υποβάλλετε νέα πρόταση για την ε, αποθήκευση δεδομένων ε, ή ε, θα διευρύνετε την συλλογή δεδομένων των επιβατών αεροπορικών εταιριών. Πρόεδρος, κύριε Ιωάννης, έχετε το λόγο. Κύριε Κέρνερ, συμφωνώ μαζί σας σε πολλά πράγματα. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τη συνεργασία τους με τη Europol εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως απάντησα και σε προηγούμενη ερώτηση, το πιο επίγον νομίζω είναι να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε αμοιβαία εμπιστοσύνη, χρειαζόμαστε αστυνομικές δυνάμεις που να συνεργάζονται πιο στενά μεταξύ τους και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε πολλές δυνατότητες τι οποίες δεν εκμεταλλευόμαστε επαρκώ ήδη σήμερα. Αυτό θα πρέπει να είναι το επικεντρό μας. Δεν αποκλείω ότι μπορεί να χρειαστούμε και άλλες προτάσεις. Νομίζω όμως ότι ε, έχουμε πολλή δουλειά όσον αφορά την εφαρμογή των όσων ήδη έχουν αποφασιστεί και να οικοδομήσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη, ώστε να συνεργαστούμε στενά στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Κυρία Κόρνερ, έχετε το λόγο. Πολύ χαίρομαι που ακούω ότι θα ε, ασχοληθείτε κυρίως με την ενίσχυση της εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών ασφαλείας. Δύο ερωτήσεις πιο συγκεκριμένες θα ήθελα να θέσω. Καταρχάς, εμπιστοσύνη όσον αφορά ε, την πρόταση για τα ηλεκτρονικά τεκμήρια. Θα προωθήσετε περαιτέρω αυτή την πρόταση και δεν πιστεύετε ότι θα είναι χρήσιμο ε, κατά την ε, επόμενη παράταση της Συμφωνίας να ζητήσετε την προηγούμενη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ και πάλι, κυρία Γιωχάνσον. Δεν κατάλαβα την τελευταία σας ερώτηση, ζητώ συγγνώμη. Εάν Εάν κατά την ε, επόμενη ανανέωση της ε, συμφωνίας ε, SWIFT με τις Ηνωμένε Πολιτείε να προβλέψετε προηγούμενη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας, κυρία Γιωχάνσον. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τεκμήρια, θα πρέπει να επανέλθω αργότερα όσον αφορά το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τις διεθνείς ε, συμφωνίες. Πολύ ευχαρίστω ε, θα ε, επιδιώξω τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωραία. Και τώρα μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τελευταίος ο συνάδελφος Πάουλο Ραντζέλ. Παρακαλώ. Κύριε Οριστήσα, Επίτροπε, καλώ ήρθατε πρώτα απ' όλα. Η ερώτησή μου είναι τελευταία, οπότε επιτρέψτε μου να τονίσω ότι μετά από την ακρόαση αυτή κινδυνεύεται να γίνεται γνωστή σαν την Επίτροπο που συστηματικά λέει θα επανέλθω, θα επανέλθω, θα επανέλθω. Το είπατε πολλές φορές σήμερα. Τα τελευταία πέντε χρόνια αναθεωρήσαμε το τοπίο της ε, Ευρώπης με προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε κενά, να δημιουργηθούν συνέργειες κτλ. Στις γραπτές σας απαντήσεις λέτε ότι θέλετε να εφαρμόσετε το νέο σύστημα. Όμως, την προηγούμενη θητεία αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά εμπόδια από κάποιες πολιτικές ε, ομάδες, μεταξύ άλλων και της δικιάς σας πολιτικής ομάδας των σοσιαλδημοκρατών. Για παράδειγμα για το VIS που καταψήφισε η ομάδα σας. Οπότε, επειδή είμαι εγώ εισηγητής για το φάκελο αυτό και επειδή έχω υπόψη μου ποια είναι η θέση των κρατών, εσείς δεσμεύεστε ότι θα θέσετε σαφή προθεσμία και συγκεκριμένον προπολογισμό για να τεθεί σε λειτουργία. Και επιπλέον πιστεύουμε ότι τα παιδιά προστατεύονται καλύτερα εάν έχουμε τα δαχτυλικά αποτυπώματα από την ηλικία των 6. Εσείς ε, θα φροντίσετε η Επιτροπή να στηρίξει αυτή την άποψη. Εσείς τώρα κυρία Γιωάννησον. Κοιτάξτε, είναι στον τριμερή διάλογο τώρα, έτσι δεν είναι. Οπότε ελπίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Δεν είμαι εγώ που θα βάλω χρονοδιάγραμμα αν δεν έχει γίνει ο τριμερής διάλογος. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα γιατί το χρειαζόμαστε. Και τώρα που λέτε ότι δεν απαντάω στις ερωτήσεις σας, μα κοιτάξτε εσείς θα αποφασίσετε, η Επιτροπή σας θα κρίνει αν εγώ απάντησα ικανοποιητικά ή όχι. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Παρακαλώ, κύριο Ραγγέλ, για άλλο ένα λεπτό. Εντάξει, το σημειώνω αυτό που λέτε. Και τώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κομμάτι του χαρτοφυλακίου σας που δεν εξετάσαμε ακόμα εδώ. Βέβαια είναι αδύνατο να τα πει κανείς όλα. Και πρόκειται για το εξή. Πώς θα υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική διάσταση της ασφάλειας. Οι πληροφορίες online, η ανάμειξη στις εκλογικές διαδικασίες είναι κάποια παραδείγματα μόνο και γι' αυτό χρειάζεται μια πιο συνεπής και συνεκτική προσέγγιση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, τα επόμενα πέντε χρόνια, τι σκοπεύετε να κάνετε ε, στο θέμα αυτό της πληροφόρησης, την ανάμειξη σε εκλογικές ε, διαδικασίες κλπ. Εσείς κύριε Γιουχάνσον. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια και ότι πρέπει να χτίσουμε και σε αυτό. Τώρα, για τις συγκεκριμένες απειλές σε βάρος των δημοκρατικών μας διαδικασιών, πρέπει να συνεργαστώ στενά και με άλλους επιτρόπους, διότι είναι ε, ζωτική σημασία να προστατεύουμε τους πολίτες μας, τις κοινωνίες μας και την δημοκρατία μας. Είναι ζωτική σημασία. Καλώ. Εδώ ολοκληρώνεται ο δεύτερος γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων και έχουμε και τελική δήλωση που είναι σύμφωνα στους κανόνες του παιχνιδιού, του εσωτερικού κανονισμού. Για να καταλάβουμε δίκαια. Αν αυτή ήταν δίκη, θα είχατε τον τελικό λόγο. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, κυρία Γιωχάνσον, έχετε λοιπόν το λόγο. Θα σας ευχαριστήσω, ευχαριστώ όλους σας για τη συνεισφορά σας που ήσασταν τόσο αποτελεσματικοί. Δείξατε μεγάλη κοινοβουλευτική πειθαρχία, περιοριστήκατε στο χρόνο που είχε προγραμματιστεί, ούτω ώστε να ασκηθεί αυτό το εγχείρημα κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με το χαρακτήρα και τα προσόντα κάθε υποψηφίου επιτρόπου και συγκεκριμένη περίπτωση της υποψηφίας επιτρόπου για εσωτερικά θέματα εσωτερικών και της κυρίας Ούλβα Γιώχανσον. Και θέλαμε αυτή η διαδικασία να λάβει χώρα με ικανοποιητικό τρόπο. Ήταν πολύ ικανοποιητικό ο τρόπος με τον οποίο διενεργήθηκε το τελευταίο δίωρο αυτή η ακρόαση δύο ώρες και ένα τέταρτο κράτη. Είναι η σειρά σας τώρα. Κυρία Γιώχανσον, η τελική σας δήλωση. Έχετε το δικαίωμα να θέσετε τέρμα σε αυτή τη συζήτηση μέσω μιας σύντομης δήλωσης, ε, όχι παραπάνω πέντε λεπτά. Έχετε ξανά το λόγο εσείς, κυρία Γιώχανσον. Σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας, που, προσπάθεια που καταβάλατε για να διασκεδάσετε τις ανησυχίες που εξεφράστησαν και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας ετέθησαν. Έχετε ξανά το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπα και στην αρχή, προσέβλεπα σε αυτή τη διαδικασία και είχα δίκιο. Είναι πάρα πολύ ικανή αυτή η Επιτροπή με πολλές αρμοδιότητες, πολλές γνώσεις σχετικά με το τι γίνεται στην πράξη σε κάθε κράτος μέλος, εκπροσωπείτε πραγματικά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ελπίζω να μπορέσω να συνεργαστώ στενά μαζί σας την επόμενη πενταετία. Προσβλέπω σε αυτό, πραγματικά. Αν βέβαια επικυρωθεί η ανάθεση των καθηκόντων μου. Είμαστε στην αρχή ενός ταξιδιού μαζί, ελπίζω, για να υλοποιήσουμε πολιτικές που είναι πολύ σημαντικές για τους πολίτες μας, για θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, διότι αυτά είναι θέματα που απασχολούν τους πολίτες μας και θεωρούν ότι πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό έχουμε μια υποχρέωση να δώσουμε αποτελέσματα. Όπως προανέφερα, είναι σαφές για μένα ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες μας εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσης Επίσης όμως πρέπει να έχουμε υπόψη και τον αντίκτυπο που έχουν οι κανόνες μας εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πάντα να ηγείται ως παράδειγμα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα ποτέ δεν θα πρέπει να είναι κάτι που το σκεφτόμαστε εκ των υστέρων. Είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Για τη μετανάστευση η φιλοδοξία μου να επιληθεί το πρόβλημα. Η κοινή μας επιτυχία θα κριθεί όχι μόνο εάν, αλλά και μέσω του πώς θα προχωρήσουμε. Θα πρέπει να βρούμε ευρωπαϊκή λύση. Άρα κοινέ λύσεις, διαχειρίσιμες, βιώσιμες, προβλέψιμες, που θα δράζονται επί των αξιών μας και των θεμελιωδών μας δικαιωμάτων. Σαφώς χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή λύση για ένα σύστημα μετανάστευσης ευρωπαϊκό που θα είναι διαχειρίσιμο Χρειαζόμαστε έρευνα και διάσωση που θα είναι κάτι πιο βιώσιμο σαν προσέγγιση. Χρειάζεται ολιστική προσέγγιση. Ένα σύμφωνο που θα προβλέπει νόμιμες ασφαλείς διόδους. Πώς θα το πετύχουμε αυτό, διαφυλάσσοντας το δικαίωμα να, ε, για υποβολή αιτήσεω ασύλου και να αξιολογείται η αίτηση γρήγορα και σωστά και ατομικά. Εκείνοι που δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να παραμείνουν θα πρέπει να επιστραφούν σύμφωνα με την νομοθεσία μας και σύμφωνα με του κοινού μας κανόνε κανόνες με αξιοπρεπή τρόπο. Αυτό συνδέεται με την αύξηση της καταπολέμησης των διακινητών. Τα συμφέροντα του παιδιού και η χρειά του φίλου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε αυτά που κάνουμε, να λαμβάνονται υπόψη σε όλε τι πολιτικέ που θεσπίζουμε. Και αυτό σα διαβεβαιώνω ότι θα το προωθήσω και το εξασφαλίσω για την ασφάλεια. Θα καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Έχουμε προχωρήσει πολύ. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει να διστάσουμε να κάνουμε και άλλα βήματα για τη βελτίωση τη ευρωπαϊκή συνεργασία και να συνεργαστούμε με περαιτέρω αύξηση εμπιστοσύνη μεταξύ των δυνάμεων επιβολή του νόμου. Όπως είπα επανειλημμένα, πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη είναι βασικό στοιχείο για τη συνεργασία στον τομέα. Εν γέννη, εύρυθμη λειτουργούσα συνεργασία στον τομέα του χαρτοφυλακίου μου είναι κρίσιμη σημασία για την εμπιστοσύνη που θα έχουν οι πολίτες μας για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όπως τόνισα προηγουμένω, συμβιβασμό και συνεργασία είναι ακρογωνία λύθη του ευρωπαϊκού τρόπου συνεργασίας. Στον τομέα του χαρτοφυλακίου μου μου ανατέθησαν πριν από τρει εβδομάδες αυτά τα θέματα και θα πρέπει να βρούμε πιο στέρεε ευρωπαϊκές λύσεις, καλύτερη συνεργασία και θα πρέπει να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη πάντα θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της συνεργασίας μας, είτε αφορά συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μεταξύ κρατών μελών ή συνεργασία με του Ευρωπαίου πολίτε. Θα πρέπει να είναι το τσιμέντο του ευρωπαϊκού οικοδομήματό μα η εμπιστοσύνη. Έτσι προτίθεμαι να προχωρήσω εάν επικυρώσετε το διορισμό μου. Και προσβλέπω στο να επανέλθω εδώ και να συνεργαστώ με αυτή την Επιτροπή που έχει πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων ε, και καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες στον τομέα. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οριστήσα, Επίτροπε Ούλβα Γιωάνσον. Θέλω εκ μέρου όλων ημών που βρισκόμαστε εδώ, αλλά και εκ μέρου ολόκληρη τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ότι εκτιμήσαμε πάρα πολύ τι προσπάθειέ σα να σταθείτε στο ύψο του χαρτοφυλακίου σας, που θα καλύψετε με το χαρακτήρα σας, και με τις ε, δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε. Ήτανε πραγματικά μία ανταλλαγή απόψεων ενθουσιώδης. Είδατε ποιο ήταν το επίπεδο της προσοχής όλων των Ευρωβουλευτών από την αρχή μέχρι το τέλος της ακρόασης αυτής. Κάτι δείχνει αυτό. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ενδιαφέρεται τόσο πολύ για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Μετανάστευση, ε, προστασία, άσυλο, όλες οι υπηρεσίες επίσης οι οποίες αποτελούν το γαλαξία της Επιτροπής μας και βέβαια για το θέμα της ασφάλειας που ήδη στην προηγούμενη ε, θητεία, την απερχόμενη, ήταν υπό την αρμοδιότητα ενός επιτρόπου. Εσείς τώρα θα καλύψετε και εσωτερικές υποθέσεις και μετανάστευση που είχε ένας επίτροπος τώρα. Οπότε η συζήτηση που κάναμε ήταν ένα καλό σημάδι. Σίγουρα δεν θα μπορούσε από μια τέτοια συζήτηση να βρεθεί λύση σε όλα τα προβλήματα. Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Το μόνο που θα είχα να προσθέσω αν μου επιτρέπετε, είναι ότι η νέα πρόεδρος, Ursula von der Leyen, υπογράμισε στην παρουσίαση που έκανε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επί τη ευκαιρία της ψηφοφορίας που είχαμε όπου ψηφίσαμε θετικά. Είπε λοιπόν τότε ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε για να ενισχύσει τις ε, εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας πρωτοβουλίας από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι νομοθετικό σώμα και η Επιτροπή μας πρέπει να είναι μια πραγματικά νομοθετική Επιτροπή και να μπορεί να έχει λόγο όχι μόνο στα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και που θα γίνουν ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και να δίνεται συνέχεια και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όπως θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ήταν μια έκθεση πρωτοβουλίας που είχα εγώ την τιμή να είμαι εισηγητής για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει ευρείες αρμοδιότητες. και βλέπετε ότι συμμετέχει σε ακροάσεις 8 οριστέντων επιτρόπων η Επιτροπή Λίμπε. είτε ω κύριε επιτροπή, είτε ω συνδεδεμένη, είτε προσκεκλημένη, σε ακροάσεις 8 επιτρόπων. Ενώ ένα είναι το χαρτοφυλάκιο το οποίο πλήρως και αποκλειστικά είναι αρμοδιότητα της ε, δικιάς μας Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Γι' αυτό και δεν μοιραστήκαμε την ακρόαση αυτή με καμιά άλλη επιτροπή. Γιατί ακριβώς το χαρτοφυλάκιό σας αντιστοιχεί απόλυτα με τις δικές μας αρμοδιότητες και γι' αυτό και είδατε τόσο ενθουσιασμό και τόση ενέργεια και τόση συμμετοχή και εμπλοκή των Ευρωβουλευτών στη συζήτηση. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι όσον αφορά την αξιολόγηση, οι συντονιστές θα συναντηθούν σήμερα αργότερα στις 7. Το που ακριβώς θα ανακοινωθεί στους ε, συντονιστές για να βρεθούμε και να εξολογήσουμε την ακρόαση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Γιωχάνσον. Λήξη της συνεδρίασης.